Right, colleagues, we're going to make a start because colleagues, everyone can take their seats. We can make a start. Συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα στην ημερήσια διαταξή, όλα σημαντικά. Και δεν θέλουμε να χασομεράμε. Να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Σημείο 2. Έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη τη συνεδρία όπω έχει υποβληθεί. Τρία ανακοινώσει του Προέδρου. Δεν έχω καμία ανακοίνωση. Έχω πει ψηφοφορία τη 11.30 βέβαια. Ελπίζω να είναι εδώ οι συνάδελφοι στι 11.30 για ψηφοφορία. Ενημερώστε και όσοι είστε εδώ τι πολιτικέ ομάδε. Σημείο 4. Ανακοινώσει τη Επιτροπή. Είναι εδώ η Επιτροπή. Α, ωραία. Έχετε τίποτα ανακοινώσεις. Ναι, παρακαλώ. Γιωβάνα Παύλικ. Εσείς είστε. Ναι, εγώ είμαι. Καλημέρα σας. Συντονίστρια από την DG Τεύκο e για τη σχέση με το Κοινοβούλιο. Μια σύντομη ανακοίνωση για σας. Ο κύριος Φερνάντο Φρυτόρο Ντεμαερών, ε, ο διευθυντής της ε, DigiDevco, αφήνει το Μάρτιο την ε, διευθυνσή μας. Έχει προσκληθεί από την Πορτοκαλική Προεδρία να αναλάβει τη θέση την διεύθυνση της ομάδας του γραφείου του Προέδρου της Πορτοκαλικής Δημοκρατίας. Θα δούμε ποιο θα διαδεχθεί τον κύριο Φορτουόζο ω διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ, αλλά θα σα ενημερώσουμε καιρό. Ευχαριστούμε. Ε, πολύ σημαντική πληροφορία. Πρέπει να το έχω πει και στου συντονιστέ προηγουμένω. Και ήταν γνωστό την περασμένη εβδομάδα. Λυπούμαστε ιδιαίτερα που φεύγει. Αλλά είναι μεγάλη τιμή ε, να τον ανακαλούν στη χώρα του για να αναλάβει τη διοίκηση ε, αυτού του γραφείου. Πριν φύγει, ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και την ευκαιρία να τον ευχαριστήσουμε αυτοπροσώπως στην Επιτροπή μα. Ελπίζουμε να τον δούμε λοιπόν να τον ευχαριστήσουμε για τη δουλειά που έχει κάνει για την Επιτροπή στην ΤΕΒΕ εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο για την ΤΕΒΕ. Θέλουμε λοιπόν να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας. Και ελπίζουμε να τον δούμε και να έχουμε την αντικατάστασή του στο μέλλον με εξίσου έστω ε, επιτυχημένο τρόπο. Σημείο 5. Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμω μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, αντίδραση στην ανακοίνωση της Επιτροπής Trade for All για μια νέα πολιτική για την αναπτύξη και τις επενδύσεις ε, από πέρσι τον Οκτώβριο. Η ανακοίνωση, πολύ σημαντικό νέο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι ξέρουμε ότι χωρίς το εμπόριο και τις επενδύσεις δεν μπορεί κανείς να έχει ούτε οικονομία ούτε ανάπτυξη. Η νέα αυτή πρόταση περιλαμβάνει και πτυχέ. Οπότε να ακούσουμε τον κύριο Ζαχραντήλα από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Έχετε κάτι διαδικαστικό να πείτε, κύριε Γκέρεντ. Σας είχα αποστείλει ένα ερώτημα, Πρόεδρε, και θέλω να το θέσω στην Επιτροπή. Κανονικά, ε, Μπορούμε να το κάνουμε αυτό στην αρχή της ε, συνόδου. Έχετε μία ερώτηση, αλλά αφορά ένα σημείο της ατζέντα στο τέλος της ε, συνεδρίασης. Οι ερωτήσεις ε, προς την Κομισιόν υποβάλλονται γραπτός όμως κανονικά. Έχετε μία ερώτηση η οποία έχει υποβληθεί και γραπτός. Σωστό. Για το σημείο 19. Ίσως δεν είναι έτοιμοι αυτοί οι εκπρόσωποι της Κομισιόν να απαντήσουν ερωτήσεις για το ερώτημα 19. Ε, εδώ φτάνουμε μέχρι το 9 ε, ή 10 σημείο. Ε, ζητώ συγγνώμη, νόμιζα ότι θα μπορούσα να υποβάλω ε, ερωτήσεις ε, στην αρχή της συνεδρίασης. Και ότι στην αρχή της συνεδρίασης υποβάλλονται ερωτήσεις. όχι, όχι, λέει η Πρόεδρος, μέχρι το 9 ή 10 σημείο θα φτάσουμε το πρωί. Κύριε Ζαχραντή, έχετε την, το λόγο για να, να παρουσιάσετε το θέμα σας. Ε, χαίρομαι που είμαι υπεύθυνο για αυτή την γνωμοδότηση, γιατί είμαι και τακτικό μέλος της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Οπότε είναι καλό από αυτήν την άποψη, γιατί συνδυάζω και τα δύο και μπορώ να βρω μια ισορροπία ανάμεσα στην ε, αναπτυξιακή ατζέντα και στην ε, εμπορική ατζέντα. Υπάρχει ένα σημείο για τις νέες προοπτικές, τις καινοτόμες στρατηγικές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ετοίμασα ένα σχέδιο γνωμοδότηση ευσύνοπτο, 7 σημεία. Δεν νομίζω ότι είναι ένα πράγμα αυτό που αφορά αποκλειστικά το εμπόριο, αλλά τονίζω τη σημασία του εμπορίου. Και με δύο λόγια να σας πω τι μπορείτε να βρείτε στο σχέδιο γνωμοδότησής μου. Τονίζω το ανοιχτό εμπόριο ως απομηχανή για την ανάπτυξη. Τονίζω τη σημασία της συνεισφοράς ε, της εμπορικής πολιτικής στην ε, βιώσιμη και αηφόρα ανάπτυξη. Επίσης, ε, καλωσορίζω το αποτέλεσμα της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι και κυρίως στον τομέα της γεωργίας. Τονίζω το σημαντικό ρόλο ε, τη βοήθεια για το εμπόριο, στη δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα του εμπορίου, στη τεχνική βοήθεια τη πολιτική επιχειρηματική στήριξη των ΙΜΕ, οι, οι συμφωνίε οικονομική εταιρικής σχέσης αποτελούν σημαντικό εργαλείο για να μειώσουμε μακροπρόθεσμα τη φτώχεια και τέλος τονίζω ότι η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες και ότι είναι απαραίτητο να την καταπολεμήσουμε να ακούσω υποδείξεις, προτάσεις με χαρά ή τροπολογίες από τους συναδέλφους και είμαι έτοιμος βεβαίως να συζητήσω τα σημεία αυτά ούτω ώστε να συμφωνήσουμε. Αυτά εν είδη εισαγωγής. Δεν θέλω να μακρηγορήσω πέραν όλων αυτών που είπα και περιμένω προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ο Πολ Ρούμπικ από το ΕΛΚ είναι ο πρώτος ομιλητής. Καταρχά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ζαχράτη γιατί αυτό το θέμα για μας θα είναι πολύ σημαντικό ε, στο μέλλον. Όπως ε, γνωρίζουμε, κάθε φορά που υπάρχει μια διάσκεψη, όχι μόνο ε, για την παραγωγή, αλλά έχει, έχει να κάνει και με την κατανάλωση. Άρα η παραγωγή, η κατανάλωση, οι επενδύσεις ε, είναι τα θέματα τα οποία ε, μπορούν να φέρουν ευημερία και θέσεις εργασίας. Άρα το πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το χωρίσουμε. Και η πρόσβαση στην αγορά για τις λιγότερο αναπτυγμένες ε, χώρες ε, σε περιοχές όπου η Ευρώπη ε, είναι η μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, που είναι η μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη του κόσμου, είναι πολύ σημαντική. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε προσφορά προϊόντων και να υπάρχει και μια συμμετοχή των, ε, στην αγορά εργασίας. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει και με τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ για τις νέες τεχνολογίες συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ψηφιακό εμπόριο. Αυτό στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί μια νέα ευκαιρία γιατί μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους στις αγορές και με αυτόν τον τρόπο. Επίσης έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι υποδομές σε αυτές τις χώρες θα πρέπει να ενισχυθούν, ας πούμε, η ηλεκτροδότηση. Για να μπορεί κανείς να κάνει ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να έχει καλύτερο δίκτυο ηλεκτρισμού και με ανανεώσιμες πηγές όπως φωτοβολταϊκά. Με αυτόν τον τρόπο ε, θα δημιουργηθεί η βάση για να υπάρχει παραγωγή και ανταγωνισμός ε, ε, που θα οδηγήσουν σε ευημερία. Πέραν τούτου είναι ξεκάθαρο φυσικά ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι για μας πάρα πολύ σημαντική και πρέπει οι σχετικοί θεσμοί στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες ε, να σταθεροποιηθούν, να μην υπάρχει διαφθορά, έτσι ώστε να αποφεύγουμε ε, τα εμπόδια για την ευημερία με το Trade Facilitation και ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να προοδεύσουν και είναι σημαντικό αυτό. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσουμε τα προγράμματα που έχουμε για τις ασθενείς περιοχές να τα επεκτείνουμε ίσως, να σκεφτούμε αν μπορούν να πάνε και στις λιγότερο ανεπτυγμένες ε, περιοχές και χώρες. Έχουμε, ας πούμε, το Εράσμους για τους νέους επιχειρηματίες. Ε, θα μπορούσαμε ε, να το προωθήσουμε και θα ήταν πολύ καλή ευκαιρία για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί πρέπει να κάνει πολλή δουλειά. Και αυτή η έκθεση είναι πραγματικά επαγγελματική και έχουμε κάνει με αυτήν ένα μεγάλο βήμα προς αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πέδρο Σίλβε Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συγκητή για το σχέδιο έκθεσης και για την προθυμία του να συνεργαστούμε επικοδομητικά. Σε αυτή την παρέμβαση της Επιτροπής για την Ανάπτυξη που μας φαίνεται σημαντική. Μιλάμε για ένα θέμα κέριο για να υπάρχει συνοχή στις πολιτικές ανάπτυξης. Μιλάμε πολύ για την αρχή αυτή, αλλά εδώ όλος ιδιαιτέρως είναι πολύ κέρια η αρχή αυτή όταν μιλάμε για την εμπορική στρατηγική της Ένωσης. Δεν θέλω απλώς να εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Θα ήθελα να αναγνωρίσω τη στρατηγική που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Trade for all περιέχει ε, μηνύματα θετικά, αρκετά θετικά, ως προς τη συμπερίληψη της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής και της επενδυτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι και πολύ θετικές σημείες που γίνονται στην πολιτική που θα βασίζεται σε αξίες που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση των δικαιωμάτων και γενικότερα το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και του δικαίου εμπορίου, του fair trade. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η Επιτροπή σκοπεύει να εκπονήσει μελέτη, λεπτομερή μελέτη των συνεπειών των εμπορικών μας συμφωνιών στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και παράλληλα την ε, συμφωνία να υπάρξουν ρήτρε για την καταπολέμηση της διαφθοράς της εμπορικής συμφωνίας. Κάτι που είναι και αυτό σημαντικό. Το πλέον σημαντικό βέβαια είναι ότι η Επιτροπή συσχετίζει και ε, φροντίζει να υπάρχει συνέπεια των λόγων με τις πράξεις και βεβαίως θα πρέπει να φροντίσει στην εμπορική μας πολιτική όντως να επιδιώκεται η, πολιτική, ανάπτυξη. Από δική μου πλευρά και για την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, σε ένα πνεύμα επικοδομητική συνεργασία, θα προτείνουμε τροπολογίε στον εισηγητή για τη γνωμοδότηση τη επιτροπή μας ε, που συζητάμε. Σε πρώτη φάση νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε όχι απλώς την συμπερίληψη σφαιρικότερων ε, κεφαλαίων για την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά να δώσουμε έμφαση και στις επενδύσεις και επίσης ισχυρή έκφραση στα κεφάλαια που εκφράζουν, που καθορίζουν το σύστημα υλοποίησης και εφαρμογής της θεωρίας των προηγούμενων κεφαλαίων. Έχουμε δει ότι ως τώρα η Επιτροπή δεν είναι πάντοτε συνεπής και πιστή σε ένα ανώτερο πρότυπο για την ε, υλοποίηση των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη τη εμπορική συμφωνία. Κάποιε περιπτώσει τι βλέπουμε σε, χώρες που σε συμφωνίε που έχουν συναυθεί με αφρικανικέ χώρε, αλλά έχουμε δει να προκύπτουν και καταστάσει όπου υπάρχει οπισθοχώρηση, η παναχώρηση του επίπεδου και του ε, προτύπου που ισχύει για την επίτευξη των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε λοιπόν εκεί να υπάρχει μια ισχυρότερη έκφραση, να δοθεί μεγαλύτερη αξία και σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και τα εργασιακά στην ισότητα των φύλων και στην προστασία του καταναλωτού. Έπειτα, κατά δεύτερον, στις ε, υποδομές για την παρακολούθηση υλοποίησης των συμφωνιών, γιατί θα πρέπει αυτές να είναι λειτουργικές και να δίνεται αξία στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Και αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί στην έκθεση της Επιτροπής μας. Κατά τρίτον, Νομίζω σημαντικό είναι να ζητηθεί να υπάρχει διάλογος και ευρύες διαβουλεύσεις οι οποίοι, οι οποίοι, τα οποία μάλλον να φροντίζουν για τη συμμετοχή, να απαιτούν τη συμμετοχή των χωρών της ΑΚΕ και για το τι θα γίνει μετά τη συμφωνία της Κοτονού. Ήδη μας έχει απασχολήσει και στην Επιτροπή μας και στην επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το τι θα γίνει για το διάστημα αφού εκπνεύσει η Συμφωνία Κοτονού και αυτό θα επηρεάσει και την εμπορική μας πολιτική. Τέλος, πρέπει να οριστεί μια σχέση συνεργασίας, μάλλον μια, ένα συνδυασμός όλων μας των εμπορικών πολιτικών για να συνδράμουμε τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών προκειμένου η εσωτερική προστιθέμενη αξία των οικονομιών τους να ευνοηθεί και έτσι να εκμεταλλευτούν το δυναμικό ανάπτυξης που διαθέτουν. Αυτή είναι η γενική προσανατολισμή των τροπολογιών που σκοπεύω να υποβάλω με, ε, μέσα σε ένα επικοδομητικό πνεύμα προκειμένου να προκύψει μια συγκροτημένη θέση της Επιτροπής μας για την εμπορική πολιτική της Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριο Γκέρεντς. Euh, Ευχαριστώ τον εισηγητή τον κύριο Ζαχαντήλ. Στην παράγραφο 2 των ε, υποδείξεων του λέει ότι είναι σημαντική αυτή η εμπορική πολιτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και υπενθυμίζει τους στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης που έχει πολλούς στόχους ε, συμπεριλαμβανομένου και του εμπορίου σε μία σειρά αποδράσεις. Είναι η πιο σημαντική ε, παράγραφος. Έχουμε δύο διασκέψεις Νέα Υόρκη και Παρίσι, όπου ελήφθησαν πολύ σημαντικές δεσμεύσεις και κυρίως ε, δεσμεύσεις που μπορούμε να επαληθεύσουμε κυρίως για τη διάσκεψη στο Παρίσι και νομίζω ότι δεν μπορούμε να τις αγνοούμε πια αυτές τις διασκέψεις που λες και δεν έχουν γίνει δηλαδή ποτέ. Δύο σημεία ανάπτυξη λοιπόν. Ε, εκπαίδευση, υγεία, εργασία, εκεί ε, διατροφή και το εμπόριο δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν μπορεί να... Δεν μπορούμε να το αποδώσουμε όλες τις αρετές και όλα τα δεινά. Είναι μία από τις πολιτικές που υπάρχουν. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής θα πρέπει να ασχοληθούμε με το αν το εμπόριο μπορεί να έχει ε, παράπλευρες δευτερογενείς επιπτώσεις στην εκπαίδευση, στην υγεία, στη διατροφή κτλ. Αθέλητες. Στα πλαίσια της νομοδότησης Νόιζερ για το ΕΚΟΒΑΣ, την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με την ΕΚΟΒΑΣ, έχουμε διατυπώσει κάποια ερωτήματα, κυρίως να δούμε ποια θα είναι η επίπτωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης στην διατροφική ασφάλεια στη ζώνη της κοινότητας των δυτικοαφρικανικών χωρών. Είναι σημαντικό το ερώτημα και πρέπει να δώσουμε απάντηση, ακόμα και αν είναι δύσκολο πολύ σωστά πρέπει να πούμε ότι το εμπόριο δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Παρόλα αυτά μπορεί να αντισταθμίσει κάποιες προσπάθειες που γίνονται σε άλλους τομείς. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και νομίζω ότι με το επίπεδο επιστήμης που έχουμε σήμερα, οικονομικής επιστήμης, δυνατότητα οικονομική ανάπτυξης που έχουμε σήμερα, θα πρέπει να τολμήσουμε να ζητήσουμε να δοθεί μια απάντηση από αυτούς που διαπραγματεύτηκαν ή που είναι επιφορτισμένοι διαπραγματευτές. Επομένως, το ερώτημά μου απευθύνεται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Μαρία Χόιμπου. Ευχαριστώ πολύ. Από την πλευρά των Πρασίνων να ευχαριστήσω για το σχέδιο αυτής της έκθεσης. Λυπάμαι λίγο που οι πιθανοί κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης του εμπορίου δεν έχουν αναφερθεί επαρκώς. Ίσως θα πρέπει να τα βάλουμε. Η απελευθέρωση του εμπορίου δεν λειτουργεί αυτόματα ως πάταξη της φτώχειας. Δεν είναι ένας αυτοματισμός. Δεν είναι ένα θαυματουργό όπλο και αυτό αναφέρεται σε πάρα πολλά σημεία, ότι οι χώρες που έχουν απελευθερώσει το εμπόριό τους ε, άνοιξαν σιγά σιγά την οικονομία τους σε συνδυασμό με τις δικές τους ικανότητες. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη γιατί έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες αγορές. Επίσης, Ε, έχει να κάνει και με μια ε, συμφωνία για τις επενδύσεις ε, που μιλάμε πλέον για δεσμευτικούς κανόνες και για μηχανισμούς βοήθειας. Και αυτά τα σημεία πρέπει να αναφερθούν. Η κοινωνική εταιρική ευθύνη στην, σε όλη την αλυσίδα παραγωγής μέσα από την πολιτική επενδύσεων ενισχύεται και ε, φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη εδώ δεν μπορούν να μιλήσουν εθελοντικά. Πρέπει να έχουν ε, οπωσδήποτε ε, σε υποχρεωτικό επίπεδο την υποχρέωση της δέουσας επιμέλειας και αυτό πρέπει να το δούμε και σε επίπεδο ομίλων, γιατί εδώ χρειαζόμαστε αυτή την υποχρεωτική προσπάθεια, την υποχρέωση ενέργειας για τις ε, βέλτιστες ε, ε, ενέργειες. Επίσης για την συμφωνία για τις επενδύσεις έχουμε να κάνουμε με πρόσβαση στη χρήση της γης. Αυτά πρέπει να τα μετρήσουμε λίγο και να δούμε και ποιες είναι οι επιπτώσεις. Να υπάρχει μια ενημέρωση των επιπτώσεων της συμφωνίας με τη Δυτική Αφρική που δεν έχει γίνει. Επίσης πολύ σημαντικό για τις νέες στρατηγικές εμπορίου είναι ο πολιτικός χώρος και τα περιθώρια που έχουν οι χώρες εταίροι. Πρέπει αυτά να τα σεβόμαστε και πρέπει να επικεντρωθούμε στην πάταξη της φτώχειας και της ανισότητας για να μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει η βιώσιμη ανάπτυξη, να υπάρχει μια κυριαρχία ως προς τα τρόφιμα και την ε, διατροφή. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα, κάνουμε, τα προσθέτουμε μέσα από τις τροπολογίες μας και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε μια θετική έκθεση και να έχουμε και επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μαρία. Δεν ξέρω, εφόσον δεν υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει το λόγο, να κάνω η ίδια κάποια σχόλια. Νομίζω ότι η νέα στρατηγική της Επιτροπής για το εμπόριο είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Εξετάζει πολύ περισσότερο τα θέματα της ανάπτυξης, της βιωσιμότητας, αναφέρει τις ε, συμβάσεις του ILO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας χαιρετίζω αυτό που γράφει ο εισηγητή στην παράγραφο 5 ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τι μικρέ επιχειρήσει και τι εταιρείε τη αναπτυσσόμενες χώρε για να μπορέσουν να είναι σε θέση να εμπορεύονται, όχι μόνο με εμά. Όταν μιλάμε για το εμπόριο συνήθω σκεφτόμαστε το εμπόριο βορανότου, όμως ε, πολλέ φορέ, σε χώρε όπω στην Κένια που ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα σημαντικό είναι και το κοινοτικό εμπόριο, το εμπόριο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό λοιπόν σε κάποιες χώρες της Αφρικής που ευτυχώς αρχίζουν να ανοίγονται. Να πω κάτι και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντική και χαιρετίζω το, το κεφάλαιο 4 του νέου γράφου της Κομισιόν. Θα καταθέσω μάλλον μόνο μία σύντομη τροπολογία. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό αυτό το κομμάτι και για την αναφορά στις βιώσιμες αλυσίδες τροφοδοσίας. Στο σημείο 2.4 του εγγράφου μιλάνε για την ε, προώθηση του δίκαιου εμπορίου και του ηθικού εμπορίου. Το fair trade, το, ηθικό το δίκαιο εμπόριο, είναι ένα μικρό κομμάτι του παγκόσμιου εμπορίου, όμως δίνει ένα παράδειγμα για το πώς το εμπόριο επηρεάζει τη ζωή των παραγωγών στις χώρες. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου ε, είχε μεγάλη δέσμευση ως προς αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα το συνεχίσει και η Ολλανδική Προεδρία. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν για την πρόταση της Κομισιόν να υποστηρίξει τους παραγωγούς του Fair Trade στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις ε, οργανώσεις της χώρας μας που ασχολούνται με το δίκαιο εμπόριο. Είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε για τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας σε αυτό το τομέα. Όλη αυτή η παράγραφος λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Και πραγματικά σας παρατρύνω να διαβάσετε αυτό το σημείο. Αυτό το έγγραφο είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ένα βήμα μπροστά ε, ως προς τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει το διεθνές της εμπόριο. Δεν ζητάει κάποιος άλλο το λόγο από ό,τι βλέπω. Έχουμε από την Κομισιόν τον κύριο Βόλπακ, από τη Γενική Διεύθυνση Trade και από την Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ ο κύριο Τζόρτζη. Ε, πείτε το όνομά σας. Ιαν Βόλβαν, ε, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Με χαρά πάντα έρχομαι στο Κοινοβούλιο, ιδίω όταν ε, ένα έγγραφο που θα ετοιμάσουμε ε, εγκομιάζεται τόσο πολύ από εσά και το Κοινοβούλιο και εσά, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα τώρα, σε σχέση με τη συζήτηση που έγινε χθε για το έγγραφο εργασία στην Επιτροπή ΙΝΤΑ. Όπω είπαν και πολλοί ευρωβουλευτέ, ε, το κείμενο προσπαθεί να αναγνωρίζει το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητιέται η εμπορική πολιτική. Ε, μάθαμε πολύ για αυτά τα πράγματα, κυρίω από τις δραστηριότητε του Κοινοβουλίου, ε, στα πλαίσια τη ευρύτερη συζήτηση που γίνεται. Δεύτερον, προσπαθούμε να βρούμε τρόπου για να εμπλακούν όχι μόνο άνθρωποι και να επηρεάσουν την πολιτική, αλλά για να την εφαρμόσουν κιόλα, όπω ακριβώ ε, είπε και η πρόεδρο. Σε σχέση με αυτό τώρα, άκουσα πολύ προσεκτικά τις παρατηρήσεις του κυρίου Ζαραχίλ, Ζαραντήλ, του εισηγητή, που βασίζεται στη, στον άξονα συζητήσεων που έκανε και η ίντα και στην ίδια την ανακοίνωση της Επιτροπής. Δεν θέλω να διατρέξω όλα τα σημεία, αλλά ε, άκουσα αυτά που είπε για το, τη βοήθεια για το εμπόριο, για τη διαφθορά, και το αποτέλεσμα του Ναϊρόμπι θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ε, στη δουλειά που κάνουμε, γιατί κάποια από τα έγγραφα ε, στην αλυσίδα παραγωγής ε, εκπονήθηκαν πριν από το Ναϊρόμπι και πριν εφαρμοστεί το Ναϊρόμπι κυρίως. Αυτό καλύπτει και πολλά από τα σημεία του κυρίου Ρούμπικ, όλα αυτά που είπα δηλαδή. Σε σχέση με τις Πατρίσει Περέιρα, η αξία είναι η βασική λέξη που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε στην ανακοίνωσή μας και η δουλειά που κάνετε για τις ομάδες παρακολούθησης ε, εντάσσονται στην αξία και στην προσπάθεια εφαρμογής που κάνουμε. Ε, για αυτό που είπε ο κύριος Γκέρεντς τώρα. Σελίδα 25, σας παραπέμπω. Ε, σελίδα 25 του αγγλικού κειμένου ε, το πρώτο, η πρώτη παύλα λέει ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει να δουλεύει με τους Αφρικανούς, ούτως ώστε να εξασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή ε, με ισχυρούς θεσμούς, ε, δομές και διαδικασίες για να ε, ενισχυστεί η καλή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου. Ε, προσπαθούμε δηλαδή να εφαρμόσουμε τις εμπορικές συμφωνίες με σοβαρότητα. Είναι δύσκολο ούτως ή άλλως να τις συμφωνήσουμε και αυτή τη στιγμή συμφωνηθούν η εφαρμογή είναι κάτι που μας απασχολεί θέλουμε να γίνει καλά και ελπίζουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει η DG Trade ε, βασίζεται σε ένα μοντέλο ε, εμπορικού τύπου. Προσπαθούμε δηλαδή να συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις ε, και στον αναπτυξιακό τομέα ε, πάλι προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τις τρίτες χώρες, με τους μη κυβερνητικού οργανισμούς με σοβαρότητα. Σας ευχαριστώ για τα κοπλιμέντα επίσης, τα καλά σας λόγια για το κεφάλαιο 4. Ε, από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, ο κύριος Κότσι, ε, σύντομα, σύντομα, μια και ο συνάδελφος είπε τα πιο βασικά. Δύο-τρία σχόλια θέλω να κάνω. Πρώτον, το εμπόριο και η ανάπτυξη ήταν τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής επί καιρό. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι πριν από τρία-τέσσερα χρόνια είχαμε δύο ε, διαφορετικά έγγραφα πολιτικής, ένα για την εμπορική και το άλλο για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Και εδώ πήγαμε ένα βήμα παραπέρα. Τονίζουμε την αλληλοσύνδεση μεταξύ των δύο. Επομένως, ε, χαίρομαι που εκτιμάτε την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Εν συνεχεία, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, ακούστηκαν σήμερα από διάφορους ευρωβουλευτές. Υποστηρίζω την συμπερίληψη κάποιων ε, αναφορών σε σημαντικές πολιτικές που θα πρέπει να είναι συνεπείς με την εμπορική πολιτική. Αλλά να τονίσω επίσης ότι αυτές οι πολιτικές αναφέρονται ήδη στην ανακοινωσή μας. Φερρυπίν, η εκπαίδευση, η υγεία, οι κανονιστικές πτυχές, ε, κλιματική αλλαγή, ε, ανθρώπινα δικαιώματα, εργατικά δικαιώματα, Κάνα πρόβλημα να μπουν στην γνωμοδότηση Επιτροπής, απλώς σας ευχαριστούμε την προσοχή ότι αναφέρονται όλα αυτά τα σημεία στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Αν λοιπόν υπάρχει τροπολογία προς αυτήν την κατεύθυνση, θα ήταν πολύ εύκολο νομίζω να βρούμε τη βάση, να βρείτε τη βάση τέλος πάντων στο έγγραφο της Επιτροπής. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Πάμε πάλι στον εισηγητή. Κυρία Τζαχαντήλ. Ναι, Πρόεδρε, δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Πρέπει να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις κέρυες παρατηρήσεις τους. Συμφωνώ με τις περισσότερες για να μην πω όλες. Με τις περισσότερες πάντως, ναι. Και θα προσπαθήσουμε να βρούμε αμοιβαίως αποδεκτούς τρόπους για να γίνει το σχέδιο αυτογνωμοδότησης ε, όπως θα το θέλαμε. Ε, απλώς μια συγκεκριμένη ε, σημεία παρατηρήσε για τη συμφωνία με το Βιετνάμ, διότι είμαι διαρκής εισηγητής για την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τη, μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Βιετνάμ. Νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να υπάρχει συνδυασμό σε μια χώρα που θεωρήθηκε πολύ φτωχή για σύστημα διεθνού εμπορίου Πώς μπορεί λοιπόν με μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου να αναπτυχθεί και μέσα σε δύο δεκαετίες να γίνει μια χώρα μέσω εισουδήματος. Νομίζω το ανέφερα αυτό. Και καλό θα ήταν να, να ακολουθήσουμε αυτή την προτροπή και να υπάρξει σχετική προπολογία. Αυτές είναι οι δικές μου παρατηρήσεις σχετικά και προσδοκώ τη συνέχιση της συνεργασίας με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ που προθεσμία για την υποβολή των απολογιών αύριο στις 6 το απόγευμα. Δεν έχετε πολύ χρόνο για την υποβολή τους, αλλά παρακαλώ πιαστείτε για να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Ίντα Εγκαίρος. Ευχαριστούμε πολύ τον συζητητή. Είναι πολύτιμη συμβολή σα και από τη δική μα επιτροπή μπορείτε να προσθέσετε τι δικέ μα τροπολογίε τι υπόλοιπε. Τώρα σημείο 6. Ένα άλλο σημείο εξίσου σημαντικό σε αυτή τη φάση. Ταμείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αφρική. Η συνέπειε για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια. Συζητούμε χωρί κείμενο σήμερα. Γιατί έτσι κι αλλιώ θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων αφού ο κύριο Κοράο μας κάνει τη βασική του σύγχυση σήμερα και αρχίσει να συντάσσει την έκθεση. Αργότερα. Είναι ένα θέμα ευαίσθητο. Με πολλές ε, πτυχές και προεκτάσεις του αποπλεγισμού, δημοσιονομικές, Είμαστε λοιπόν επιτροπή που ε, συμμετέχουμε στην όλη διαδικασία για το θέμα αυτό. Αύριο έτσι αλλιώς θα μιλήσουμε για τα θέματα της μετανάστευσης στις 10 και το θέμα της Αφρικής. Προφανώς θα προκύψει στις συζητήσεις, εγώ ίδια θα έχω συζητήσει με προσώπους των χωρών της Αφρικής. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είναι μείζωνα τα ζητήματα που δείχνονται σήμερα και χωρίς καθυστερήσει να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Κοράο. το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική υπογράφηκε από τον πρόεδρο Juncker της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 25 ε, κράτη-μέλη, συν Νορβηγία και Ελβετία και ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου του 2015 στην συνοκορυφή της Βαλέτας με τους Αφρικανούς εταίρους. Ο βασικός στόχος ε, του Ταμείου είναι να βοηθήσει για να υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή και να συνεισφέρει σε καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης. Πιο συγκεκριμένα έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τις βασικές αιτίες της ε, αποσταθεροποίησης, υποχρεωτικής ε, μετακίνησης και ελαφρομετανάστευσης με ίσες οικονομικές ευκαιρίες, ε, ασφάλεια και ανάπτυξη. Το Ταμείο για την Αφρική είναι ένα εργαλείο ε, με κονδύλια από διάφορους δωρητές, ούτως ώστε να δοθεί μια γρήγορη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνθήκες επίγουσες και κρίσεις. Ε, το Ταμείο θα βοηθήσει διάφορες αφρικανικές χώρες, ε, τις πιο ευπαθείς και τις ε, κυρίως πληττόμενες από την μετανάστευση και που θα υποφεληθούν από την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι, μη επιλέξιμες χώρες αλλά που είναι όμορε μπορούν να περίπτωση να υποφεληθούν ούτω ώστε να αντιμετωπιστούν τα ε, διασυνοριακές προκλήσεις και μετανάστευση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, τους λόγους ε, της μετακίνησης, της υποχρεωτικής μετατόπισης των ανθρώπων, της μετανάστευσης κτλ. Βασίζεται σε πέντε προτεραιότητες. Πρώτον είναι ε, η το αναπτυξιακό όφελος της μετανάστευσης. Νόμη μετανάστευση και κινητικότητα, ε, προστασία κατά της λασσομετανάστευσης επιστροφή, επανεισδοχή, επανένταξη. Η Κομισιόν ε, έχει 1,8 δισεκατομμύρια ε, στη διάθεσή της και επιπλέον κονδύλια από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους δωρητές. Το Ταμείο συμπληρώνει την ε, αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, περιοχή που θα δοθούν, δηλαδή που θα φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020, ούτως ώστε να υπάρξει μία ε, συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη. Χαρακτηρίζεται από τρεις φάσεις. υπόσχεση, δέσμευση και πληρωμή. Όπως και στο προηγούμενο ταμείο, συχνά πολλές υποσχέσεις Δυστυχώ ακολουθήθηκαν από λίγε δεσμεύσει και δράσει. Το Ταμείο θέλει να χρησιμοποιήσει ε, και τα κονδύλια που δίνουν ε, τα κράτη-μέλη με μόχλευση, ούτω ώστε να αυξηθεί η συνολική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όταν τα κράτη-μέλη δεν δίνουν επαρκή αναπτυξιακή βοήθεια, 0,7% μάλιστα, το Ταμείο θα προσπαθήσει να πιέσει τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους. Τουλάχιστον το ελπίζουμε. Ε, τα κονδύλια για το Ταμείο θα έρθουν από, τις, τα 11 αναπτυξιακά ταμεία της Ένωσης ε, με συμπλήρωμα ε, για την Κεντρική και Ανατολική Αφρική. Έχουμε το αναπτυξιακό ε, εργαλείο και το το Ευρωπαϊκό Εργαλείο ε, Γειτονίας. Ε, ένα δισεκατομμύριο ε, ευρώ δίδονται, ως, ε, δίδονται επιπλέον. Θα πρέπει αυτά τα περιθώρια να διατηρηθούν, ούτω ώστε τα ταμεία, τα κονδύλια του EDF να χρησιμοποιηθούν πραγματικά για το βασικό πρωταρχικό σκοπό που είναι η ανάπτυξη. Η χρησιμοποίηση του EDF και τα αναπτυξιακά κονδύλια των κρατών μελών για τη χρηματοδότηση του Ταμείου δημιουργεί τον κίνδυνο οι πιο φτωχές χώρες να μην ε, πάρουν κονδύλια ε, παρά τη, σημαντική, ε, τη σημασία της ODA για τις λιγότερες ανεπτυγμένες χώρες. το 2014 ήταν δεύτερη χρονιά που μειώθηκε η ODA και έχουμε τα λιγότερα κονδύλια εδώ και 10 χρόνια που δίδονται στις πιο φτωχές χώρες. Δεν θα θέλαμε οι πιο φτωχέ χώρες να πληγούν ε, γιατί θα τους αφαιρεθούν τα κονδύλια ε, για να αντιμετωπιστούν ε, οι σημερινές κρίσεις. Και θα πρέπει το 0,7% του ΑΕΠ να δίδεται στην αναπτυξιακή βοήθεια και, και ένα ποσοστό το 15% του 0,7% να δίνονται σε λιγότερο αντιγμένες χώρες. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις τοπικές υπηρεσίες, την διατροφή, τη διακυβέρνηση, το ταμείο, η, η ΜΚΟ ε, και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο για να αντιμετωπίσει τι βασικέ αιτίε και την βελτίωση των τοπικών υπηρεσιών. Το Ταμείο θα ε, εστιάσει σε μικροπρογράμματα αλλά και θέματα που απασχολούν τον κόσμο για τη βελτίωση των υπηρεσιών. Η υγεία είναι βασικός τομέας για την αύξηση της ένταξης ε, και της ανάπτυξης του τοπικού πληθυσμού. Ε, αποδεικνύεται ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες ε, όταν αποκρίνονται τις ανάγκες των ευπαθών στρωμάτων του πληθυσμού μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερες υπηρεσίες στο γενικό πληθυσμό. θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για να υλοποιηθούν οι στόχοι και το Ταμείο ε, μπορεί να συμπεριλαμβάνει και κάποια στοιχεία που δεν θεωρούνται αναπτυξιακή βοήθεια. Έλεγχο των συνόρων και αύξηση της ε, ασφάλειας της χώρες. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η διαχείριση της ε, μετανάστευσης, πέρα από τη μείωση της στόχη. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, 208 ε, συγγνώμη, της τη Λισαβόνας, ο τελικός στόχος του Ταμείου είναι μείωση και η εξάλληψη της στόχιας. Το Ταμείο χρησιμοποιεί ε, τους πόρους της ODA, όμως ο μηχανισμός του Ταμείου δεν α, εστιάζεται μόνο στην ανάπτυξη. Θα πρέπει να γίνει ε, διάκριση ανάμεσα στις αναπτυξιακές δραστηριότητες και ανάμεσα στις δραστηριότητες διαχείρισης ε, της μετανάστευσης μέσα στο Ταμείο. Το να μειωθεί η ODA, ούτως ώστε ε, να χρησιμοποιούμε λιγότερα κονδύλια για την ε, καταπολέμηση της στόχης, αυτό θα υποσκάψει τους στόχους ε, ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δράσει αυτό το επίπεδο της ανάπτυξης πρέπει να έχει μια τετραπλή προσέγγιση. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις συνδεσμεύσεις της. Επίσης να υπάρχει συνολικό συνέπεια στις αναπτυξιακές της πολιτικές, ιδίως στο πώς εφαρμόζει το πνεύμα ε, των ε, συμφωνιών ΑΚΕ μετά την Κοτονού. Θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και να αποφεύγει τις αντιφάσεις. Προς στιγμήν το καταπιστευματικό ταμείο συνδυάζει τους πολιτικούς στόχους με την πολιτική ασφάλειας, την πολιτική μετανάστευσης και την πολιτική ανάπτυξη χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική. Πρέπει να υπάρχουν κριτήρια που να διέπουν τον προπολογισμό του Ταμείου και να σέβονται τι θεμελιώδει αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπ' αυτήν την έννοια, η συνεργασία για την ασφάλεια, το οργανωμένο έγκλημα και του συνοριακούς ελέγχου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ανθρωπίνα, ανθρώπινα δικαιώματα με συγκεκριμένε διατάξει για να ενισχυθεί ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου. Με ιδιαίτερη προσοχή στα γενικά δικαιώματα, τα παιδικά δικαιώματα των μειονοτήτων και άλλων ευάλωτων ομάδων. Για τους στόχους λοιπόν τώρα. Ε, εάν ε, δούμε την επικρατούσα ασάφεια στους στόχους του θερματικού ταμείου, ακόμη και την έλλειψη αλληλεγγύης και την έλλειψη συνένεση μεταξύ των καταμελών, μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τους στόχους ασφάλειας που θεωρητικά έχουν επινοηθεί για να επιδιωχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι, αλλά θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο να ε, καθορίσουμε πώ τα κονδύλια θα αξιοποιηθούν και πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρηματοδοτήσει μέσω του ε, Αφρικανικού Ταμείου το ε, θέμα αυτό. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει στοχευμένε δράσει μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Αφρικανικά κράτη στην εκταμείευση των κονδυλίων αυτών. Το, το γεγονό ότι δεν υπάρχει συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου στην οργάνωση του Ταμείου αυτού θα πρέπει να οδηγήσει σε συστηματική υποβολή εκθέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ λειτουργεί το Καταστατικό Ταμείο, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει πλήρω ω θεματοφύλακα. Το ίδιο και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρω στη φάση τη υλοποίηση. Επιπλέον, υπό την ίδια προοπτική, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στι διατάξει που θα περιέχει ο κανονισμό του Καταπιστηματικού Ταμείου, ιδίω ω προ την υλοποίηση των διατάξεων για τη δημιουργία των hot spot ε, για την μετεγκατάσταση, την επανεγκατάσταση στι διάφορε περιοχέ, τι οικονομικέ δεσμεύσει των κρατομελών και τα κατημέλη θα πρέπει να παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να υπάρχει ο σεβασμό του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικέ τη στον τομέα αυτό θα πρέπει κυρίω να αντιμετωπίσουν τα γενεσιρουγά αιτία τη μετανάστευση, προκειμένου να υπάρχει ειρήνη, σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη στι χώρε προέλευση. Και προκειμένου να διοργανωθούν νόμιμες μετανάστευση για να υπάρχει προστασία των μεταναστών και των ασύλων, αλλά και των επανώτων ομάδων και μεγαλύτερη ε, και καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων που διατίθενται ώστε η συνεργασία και η επανεισδοχή να είναι δυνατές. Um, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε για αυτή την υπέροχη εισαγωγή. Ο κύριος Βέντα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Ως και όντως εισηγητής εκ μέρους του ΕΛΚ να ευχαριστήσω τον κύριο Κοράου για τη συνεργασία ως τώρα και για τη δυνατότητα που μας δίνεται για την ανταλλαγή απόψεων. Το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική μπορεί να γίνει ένα βασικό εργαλείο που θα ενθαρρύνει τις αφρικανικές χώρες να συνεργαστούν και στο θέμα της μετανάστευσης. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η σταθερότητα και η ανάπτυξη είναι ένα σημαντικό στοιχείο και δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στο να θέλουμε να μειώσουμε την μετανάστευση. Αυτό το ταμείο πρέπει να εφαρμοστεί γρήγορα και πρέπει να γίνει γρήγορα η διανομή των κονδυλίων ε, μεταξύ των χωρών. Πρέπει να διασφαλιστεί και να γίνει γρήγορα. Τα κράτη-μέλη δίνουν πολύ λίγες πληροφορίες. Στην ουσία δεν αντικατοπτρίζουν τις δεσμεύσεις τους. Από την άλλη, οι αφρικανικές χώρες πρέπει να διασφαλίσουν ότι και αυτές τηρούν τις δεσμεύσεις τους. Και αυτό φυσικά πρέπει να συνδυάζεται και με την συνεργασία τους, το, συνεργασία τους στο θέμα υποδοχής των μεταναστών. Οι περιοχές αυτές είναι μεταξύ των πιο ασταθών στον κόσμο. Ένας από τους στόχους του Ταμείου, λοιπόν, είναι να αντιμετωπιστούν ακριβώς οι αιτίες αυτής της αστάθειας. Να τονιστεί στην ουσία η ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας για να μπορέσουν να μεγιστοποιηθούν και οι επιπτώσεις της προσπάθειας για να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή. Για την ανάπτυξη του ντόπιου δυναμικού και τη σταθερότητα ε, πρέπει ε, ό,τι είναι να γίνει να γίνει μέσα στα χρόνο διάρκειας του project. Επίσης, πρέπει να διασφαλιστούν οι αρχές της συμπληρωματικότητας. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτό. Ενρή και Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κοράου και τον συγχαίρω. Όχι μόνο για την έκθεση, αλλά και για την ευρύτατη αυτή παρουσίαση που μας έκανε και μας επιτρέπει τελικά όχι μόνο να διαβάσουμε το περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά να το αξιολογήσουμε πολιτικά. Με βάση τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Γενικά, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ ευρεία συνένεση. Ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανάπτυξης στην Αφρική με μεγαλύτερη έτσι, σοβαρότητα και φιλοδοξία και με εργαλεία όπως το καταπίστευμα αυτό που μας επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και μια μεγαλύτερη και γρηγορότερη εκτέλεση. Αυτά είναι εργαλεία πολύ καλά, αυτά να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Και θα τα πω πολύ συνοπτικά ποια είναι αυτά τα, αυτές οι προϋποθέσεις. Πρώτον, να μην υποκαθιστά άλλες πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούσαμε πριν. Δηλαδή, να μην αλλάμε, αλλάξουμε το χρήμα, δηλαδή το πάμε από τη μία τσέπη στην άλλη. Γιατί έτσι ίσως έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά δεν έχουμε αρκετή φιλοδοξία για να επιλύσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Δεύτερη προϋπόθεση είναι να μην χρησιμοποιούμε χρήμα το οποίο προορίζεται για την ανάπτυξη και να πηγαίνει σε άλλες δραστηριότητες που δεν έχουν καμία σχέση με την ανάπτυξη. Υπ' αυτή την έννοια η χρήση κονδυλίων για την προστασία πούμε, των συνόρων ή κάτι αντίστοιχο δεν νομίζω ότι κολλάνε με αυτό που εμείς ε, κατανοούμε ως ταμείο για την ανάπτυξη. Και τρίτον, το Κοινοβούλιο μέσω της ενημέρωσης θα μπορούσε να ασκήσει ένα ρόλο παρακολούθησης και ελέγχου. Να ε, ελέγχει δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα καταπιστευματικά εργαλεία. Συνοπτικά λοιπόν. Ναι, ναι στο ταμείο, αλλά, αλλά με κονδύλια επιπρόσθετα και όχι κονδύλια τα οποία έχουν, τα έχουμε πάρει από αλλού. Υπ' αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ απογοητευτική η συνεισφορά των κρατών μελών. Και επίσης ε, τα κονδύλια που θα δίδουμε θα πρέπει να πηγαίνουν για την ανάπτυξη και όχι άσχετες δραστηριότητες που δεν κολλάνε με την έννοια της ανάπτυξης. Και τρίτον, η παρακολούθηση από το Κοινοβούλιο της εφαρμογής, της εκτέλεσης των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο λοιπά, Όπως σας είπα, προφανώς ε, στηρίζω και την εστίαση και το περιεχόμενο της έκθεσης Κοράου. Ο κύριος Ντέβα. Συγχαίρω τον κύριο Κοράο για την πολύ καλή έκθεση. Τα καταπιστεύματα χρησιμοποιούνται ευρέως όταν υπάρχουν κατεπήγοντα. Για το τσουνάμι ας πούμε δείγμα του ΟΗΕ τότε για το τσουνάμι. Και η διανομή των κονδυλίων έγινε πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ διαφανώς και δόθηκαν χρήματα στους πληγέντες που έχασαν ε, και βιός και ζωές κτλ. Και, και τους αγαπημένους τους. Για πρώτη φορά, εδώ και καιρό, η διεθνής κοινότητα και τα κρατημέλη και οι λαοί μας συνδέουν τη δική τους ασφάλεια με την ευημερία και ασφάλεια των φτωχών λαών. Επί μακρόν αυτή η σχέση δεν ε, προέκυπτε έτσι. Τουλάχιστον σε εμά στην ε, Αναπτυξιακή Επιτροπή. Και υπήρχαν άνθρωποι στις ε, χώρες μας που λέγανε γιατί δίνετε όλα αυτά λεφτά στους στοχούς είμαστε οι βασίλεις. Για πρώτη φορά συνδέουν τι εξή έννοιε. ότι αν δεν δημιουργήσει ε, σταθερές γειτονίες γύρω από τη δική μας περιοχή και δεν δημιουργήσει ασφάλεια και δυναμικό για τους στοχούς στις αναπτυσσόμενε χώρες, αυτό θα γυρίσει μπούμεραν σε εμά. Υπήρχε ένα χαζό επιχείρημα που κάποιοι τους συντηρητικούς ε, χρησιμοποιούσαν ότι θα πρέπει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, ούτω ώστε να πλουτίσουν και να κάνουν εμπόριο μαζί σου, ούτω ώστε όλοι να πλουτίσουν από κοινού. Δεν είδα ποτέ αυτή τη σύνδεση, ότι οι φτωχοί που ζουν σε φοβιστερά και ανασφαλή περιβάλλοντα μπορεί να θέλουν να κάνουν κάτι γι' αυτό, πρώτον. Δεύτερον, μπορεί να πάρουν τα μπογαλάκια τους και να φύγουν όπως κάνουν τώρα εκατομμύρια ανθρώπων. Επομένως αυτή η λαμπρή ιδέα που εμείς την καταλαβαίνουμε γιατί ασχολούμαστε με τα αναπτυξιακά, μόλις πρόσφατα ε, το αντελήφθησαν οι περισσότεροι. Και η σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη και στη μαζική μετανάστευση έθνης έγινε το πιο ε, σημαντικό πολιτικό θέμα στην Ευρώπη. Έχουμε μια τεράστια ευκαιρία, Πρόεδρε, να αδράξουμε την ευκαιρία, να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στο θεματολόγιο, στην ατζέντα. Καταρχάς, να υλοποιήσουμε τους στόχους της χιλιετία αντιξιακούς στόχους της και τώρα τους στρατηγικούς αυτούς αντιξιακούς στόχους, αλλά κυρίως πραγματικά να δημιουργήσουμε δυναμικό σε αυτές τις φτωχές χώρες, ούτω ώστε να μην χρειάζεται να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί. Ή να μην χρειάζεται να εξαρτώνται από την ελλημοσύνη μας. Αλλά πραγματικά να μπορούν να δημιουργούν ε, μια βιώσιμη ζωή. Έτσι θα πρέπει να το δούμε το καταπίστευμα αυτό. Και όχι ως εμβαλωματική λύση. Ε, κάτι που κάναμε ε, στο παρελθόν με τα καταπιστεύματα. Προσπαθούσαμε έτσι σαν μπαλώμα, με μπαλώματα να διορθώσουμε κάτι κατεπήγον. Θα πρέπει αυτό το καταπίστευμα να γίνει πραγματική ατμομηχανή δημιουργία δυναμικού, ανάπτυξη για βιώσιμη ζωή. Δεν ξέρω αν οι διευθύνοντε θα έχουν αυτή την ικανότητα να το κάνουν, τα κονδύλια να το κάνουν, τη θέληση να το κάνουν αυτό ή θα είναι κάτι προσωρινό, ε, μια προσωρινή εμβαλωματική λύση σε, ένα, σε μια χένουσα πληγή. Ο κ. Γκέρεντς. Ευχαριστούμε. Ο εξεφωνήμων ε, γείτον έχει κάνει μια πολύ καλή παρουσίαση αλλά θέλω να θέσω μια ερώτηση για τα ζήτημα ουσία. Για την υποστεθέμενη αξία που μπορεί να παρουσιάζει το εργαλείο αυτό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι πρώτε τη διαβουλεύσει και στα σχολεία τη το παρουσίασε ω ευελικτότερο που θα επιτρέπει να εκταμιευθούν πιο εύκολα τα ποσά σεβόμενοι και λαμβάνοντα υπόψη του κανόνε που ισχύουν στην Επιτροπή. Οπότε είτε θα βασιστούμε στου κανόνε που, που, ισχύουν, είτε πρέπει να μου εξηγήσει κάποιο γιατί να επινοηθεί αυτό το εργαλείο. Δεύτερον, ο εισηγητή είπε ότι το καταπίστευμα σκοπό έχει να καταπολεμήσει την αστάθεια στην ε, περιοχή τη Βορειοαφρική. Τέλεια. Αλλά μετά μιλάει για παρεμβάσει στο εκπαιδευτικό σύστημα, το γενομικό, τη ασφάλεια και την, μετανάστε, την ε, μετανάστευση για να τα καταφέρουμε όλα αυτά. Για την εκπαίδευση πιστεύω ότι έχουμε τα ανάλογα εργαλεία. Και για το υγειονομικό το ίδιο. Για την ασφάλεια νομίζω εκεί έχουμε να κάνουμε με προβλήματα άκρος δύσκολα και εντελώς καινούρια. Ποιος θα διοργανώσει την ε, ε, παρέμβαση αυτή στο Μάλι λόγου χάρη έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό το Μάλι για να κάνει αυτά που πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Γαλλία πιστεύω ότι παρακολουθεί την κατάσταση εκεί. Θα πρέπει λοιπόν οι χώρε να ασχοληθούν καμιά εικοσαετία για να καταφέρουν να πετύχουν ε, να εκπληρώσουν αυτέ τι απαιτήσει. Δεν έχουν τα μέσα αυτή τη στιγμή. Και τα μέσα αυτά ε, εκεί που τα ε, βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό με την ανάπτυξη. Μετανάστευση τι μπορούμε να παρατηρήσουμε για τη μετανάστευση. μετανάστευση εντό τη ίδια γεωγραφική ζώνη, από το Μάλι στην Μπουρκίνα Φάσο, από την Γκάνα στο. Ε, ε, στην ε, ακτή του Λεφαντοστού και ούτω καθεξής. Αλλά θα δούμε αυτή την περιφερειακή μετακίνηση ε, στην ίδια γεωγραφική ζώνη ή προς τις δικές μας χώρες. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στου στόχου μα λοιπόν. Αν θέλουμε να προλάβουμε τη μετανάστευση προ τι δικέ μα χώρε, θα πρέπει βεβαίω να παρέμβουμε στο εκπαιδευτικό, υγειονομικό και στι υπόλοιπε συνιστώσει τη ανθρώπινη ανάπτυξη. Αλλά ε, κατά τρίτον πρέπει να διερωτηθώ για τα εργαλεία. Τα εργαλεία και του εταίρου. Του εταίρου που θα πρέπει να προσεγγίσουμε στον τομέα αυτό. Ποιοι είναι οι εταίροι μα. Το καταπίστευμα αυτό το Trust Fund θα απευθύνεται στα επιμέρους κράτη ή θα ανατρέξουμε, θα ψάξουμε κάποιον ε, περιφερειακό εταίρο, ε, επιτόπιο, όπως την κοινότητα των κρατών της Ανατολικής Αφρικής, της CDAO, όπως λέγεται σε σύνδεση. Έχει επιτροπές η Ένωση αυτή. Έχει οργανωθεί κατά τρόπο ώστε θεωρητικά τουλάχιστον να μπορεί να καλύψει όλε τι μεγάλε τη ανάγκε. Η ερώτηση είναι η εξή. Θα είναι αυτή ο ιδανικό ε, συνομιλητή. Και θα διερωτώ μέχρι και το εξή. Είναι ο ιδανικό συνομιλητή, οπότε πρέπει να την προσεγγίσουμε δημοσιονομικώ. Μήπως αντί να φτιάξουμε ένα καταπίστευμα που θα το χειρίζονται ένα σωρό εμπειρογνώμονες που μπορούν να μπλοκάρουν τις δυναμικές ε, σχέσεις στα πλαίσια της Επιτροπής. Μπορεί αυτό τελικά να μας κάνει να κατασπαταλήσουμε άδικα ανθρώπινους πόρους. Εμπιστευόμαστε λοιπόν μια τέτοια περιφερειακή οργάνωση όπω αυτή των κρατών τη Ανατολική Αφρική, εκεί που υπάρχουν στατικικέ εταιρικέ σχέσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ένωση ή θα την παρακάμψουμε. Νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε. Νομίζω ότι αυτή η ένωση των κρατών της Ανατολική Αφρική είναι η φωτοτυπία των όσων κάνουμε στην Ευρώπη. που εμά έχει πνευστεί και προσπαθεί να κάνει ακριβώς τα ίδια με εμά. Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση για τη σταθεροποίηση και την ειρήνη, το εργαλείο αυτό τους ενδιαφέρει τους εταιρούς μα, έτσι θα είναι η, Ένωση, η Αφρικανική Ένωση που ήδη παίρνει χρήματα από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο, ιδίω για τα peace facilities, από εμά. Αυτή θα είναι ο συνομιλητή, γιατί νομίζω ότι έχουμε όλο τη φαρέτρα των ε, απαραίτητων ε, βελών που θα πρέπει να το ξέψουμε, εάν θέλουμε να πετύχουμε του σωστού εταίρου. Και τέλος, τελευταίο σημείο, διερωτώ με, εάν είναι ένα εργαλείο που ενδιαφέρει την Επιτροπή και τον Πρόεδρο τη πραγματικά. Διότι αν δω τι γίνεται σε αυτή την Επιτροπή, εάν δω την ε, χλιαρότητα με την οποία ε, ανακοινώνουν ε, την δέσμευσή του στα κάτι μέλη, όπως τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη Βαλέτα, στην Κοινή Συνόδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικανικής Ένωσης, Ε, εδώ λοιπόν, εάν δούμε την επιπολαιότητα αυτή, ανακοινώθηκαν κάποια ποσά, αλλά δεν έχουν ακόμη ταμιευθεί. Ε, αυτά τα ποσά θα έχουν πλέον συμπερίληψη στον προπολογισμό και θα χρησιμοποιηθούν για να υπολογιστεί η συνεισφορά των κρατών μελών ως τα δημόσια τα κονδύλια προς τη δημόσια ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια. Ούτε ένα λεπτό του ευρώ δεν θα προσθεθεί. Αυτά που μπορεί να προέλθουν ως καινούρια θα είναι από την Αφηγία και την Ελβετία. Ας είμαστε λοιπόν κάπως αντικειμενικοί. Υπάρχει η θέση της ουσίας, το πρόβλημα της ουσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, πάρα πολύ κακή στις επιδόσεις, στο επίπεδο των κρατών μελών και από αυτήν την κριτική απλώς θα εξαιρέσω το Ηνωμένο Βασίλειο, όπω έφτασε στο 0,7%. Γιατί εκεί νομίζω πρέπει να αποτύσσουμε φόρο τιμή. Είναι η μόνη χώρα που κράτησε την υπόσχεσή τη και από το 2004 έχει παραμένει πιστή σε αυτή την υπόσχεση. Την υπόσταση για την αναπτυξική βοήθεια. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι δεν χρειάζεται να εφεύρουμε ένα καταπιστευματικό ταμείο εδώ πέρα γι' αυτό, ούτε νέα εργαλεία θα μπορούσαμε να ε, συγκεντρωθούμε στην ενίσχυση των υπαρχουσών δομών ή τέλο πάντων εφόσον υπάρχουν ελλείψεις αυτές να τις συμπληρώσουμε. Από αυτή την άποψη το καταπιστευματικό θα μας έδειχνε και πού ακριβώς υπάρχουν τα κοινά και οι ελλείψεις. Ευχαριστώ κυρία Χάταλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πώς Εμείς που υπερασπιζόμαστε τις αρχές της αναπτυξιακής πολιτικής και της αποτελεσματικότητας, πρέπει να είμαστε πολύ κριτικοί ως προς αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο. Είναι δύσκολο κανείς να αντιταχθεί σε αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Μάλλον, στην ουσία είναι ένας τρόπος για να δώσουμε την εντύπωση ότι παίρνουμε στα σοβαρά την μετανάστευση και ότι αντιμετωπίζουμε τις ρίζες του προβλήματος. Και έτσι να υποχρεώσουμε τις χώρες εταίρους να συνεργαστούν στο θέμα της μετανάστευσης και να μπουν σε συμφωνίες για την επιστροφή προσφύγων από τις χώρες μας. Δεν είναι λοιπόν κάτι όμορφο και ξεκάθαρο, είναι η λογική συνέπεια του πώς αντιδρούν οι πολιτικοί όταν υπάρχει κρίση. Δεν είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Και έχω μεγάλο σκεπτικισμό σχετικά με αυτή τη νέα συζήτηση για την ε, ανάπτυξη και την ασφάλεια. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς την ασφάλεια και ασφάλεια χωρίς την ανάπτυξη. Ναι, αλλά τώρα ε, αυτό που λέμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τα λίγα χρήματα που γίνονται όλο και λιγότερα στον προϋπολογισμό για την ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των προσφύγων και τις ρίζες του. Ας μην υπερβάλλουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν, και αν είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στον κόσμο, ακόμα δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τις ρίζες του προβλήματος. Οι άλλοι δωρητές ακόμα λιγότερο. Και τώρα έχει ε, εξαπλωθεί πια η φωτιά και πρέπει οι αρχές της ανάπτυξης να εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Πρέπει να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό της βοήθειας και να δοθούν τα χρήματα σε σκοπούς που δεν προωθούν την ανάπτυξη αλλά μόνο την ασφάλεια. Πρέπει σε αυτό να αντιταχθούμε. Ο εισηγητής μας επίσης ανέφερε ότι εδώ δεν εφαρμόζεται η διαδικασία της εξέτασης της, του ελέγχου. Πώς εμείς λοιπόν ε, θα μπορούμε να τα ελέγξουμε ότι, να ελέγξουμε ότι σε κάποιο βαθμό γίνονται αυτά που πρέπει. Ο, ο Ιγνάζο ανέφερε ότι η απέτηση της Επιτροπής για την αναφορά και το reporting είναι ε, ακόμα μεγαλύτερη από ότι είναι φυσιολογικά λόγω της έλλειψης ε, της εξέτασης, του δικαιώματος εξέτασης. Δεν ξέρω λοιπόν ε, αν είναι κάποιο μαγικό τρίκ αυτή τη στιγμή που όλα τα κράτη-μέλη μειώνουν τον προϋπολογισμό τους. Ε, είναι ατυχής η κατάσταση, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Οι κυβερνήσεις ζητούν να γίνουν περισσότερα, χωρίς όμως να δίνουν τα μέσα για να γίνουν περισσότερο. Και Υπουργοί ανάπτυξη στο αντίστοιχο Συμβούλιο είπαν ότι περισσότερα πρέπει να γίνουν, αλλά χωρί να συζητήσει με του υπουργού Οικονομικών δεν μπορεί να κάνεις περισσότερο. Τώρα από την ε, ε Κομισιόν, από την DG ο κύριος Πέρτς, έχετε κάποιες ερωτήσεις, κάτι να προσθέσετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεση και για το feedback από τον εισηγητή. Να δώσω και εγώ κάποιο feedback και κάποιες απαντήσεις ε, καταρχάς για να πω και να διασφαλίσω στην Επιτροπή σας ότι ο κώδικας θα, θα γίνει σεβαστό, σεβαστός ο κώδικας ΤΑΚ και ότι όλα τα θέματα που θα σχετίζονται με αυτό το ταμείο θα έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Ακόμα και αν υπάρχει διαχείριση των συνόρων και θέματα ασφαλείας, όλα αυτά θα γίνονται ε, βάσει του κώδικα για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Για την συνεισφορά των κρατών μελών, η Κομισιόν παρά μόνο να συμφωνήσει μπορεί θα επαναλάβω αυτό που υπόθηκε. Είναι μια ομοιοπαθητική και χαιρόμαστε που έχουμε πολύ περισσότερα κονδύλια τώρα. Η Κομισιόν ίσως θα πρέπει να δείξει, να καταδείξει ότι είναι δυνατό να έχουμε αποτελέσματα για να μπορέσει να πάρει περισσότερα κονδύλια. Αν γίνει αυτό λοιπόν με θετικό τρόπο και είναι επιτυχημένο το Trust Fund θα έχουμε επιπλέον κονδύλια. Επίσης αυτό το ταμείο δεν ε, είναι ένα ταμείο που είναι ταμείο ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά ταμείο ανάπτυξης. Έχει συγκεκριμένα εργαλεία, συγκεκριμένα μέσα. Ακόμα και αν υπάρχουν κάποια μοσά, ποσά που έχουν μεταφερθεί, έχουν να κάνουν με το ίδιο θέμα της ανάπτυξης. Είναι ένα Μέσω εφαρμογής. Δεν είναι χρηματοοικονομικό. Το οποίο τροφοδοτείται από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα. Αυτό που πρέπει να προάγουμε λοιπόν εδώ είναι το γεγονός ότι μπορέσαμε να δημιουργήσουμε ένα trust fund τα οποία, το οποίο θα παίρνει λεφτά από τον DCI, από την ΕΚΟ, από, το, από τους το τομείς ε, που ασχολούνται με την ανάπτυξη. Είναι ένα πιο γενικό ταμείο το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στην Αφρική, στο σύνολό τη και στη Βόρεια και στη Νότια Αφρική. Επίσης για την προστιθέμενη αξία του Trust Fund και για τους κανόνες της ευελιξίας που δόθηκαν, φυσικά θα σεβαστούμε τους κανόνες. Αυτό που σας είπα είναι ένα εργαλείο εφαρμογής και είναι πιο γρήγορη η λήψη αποφάσεων. Έχει ήδη πάει στην επιστροπή Fed το Trust Fund και μπορούμε να αποφασίζουμε βάση των αναγκών. Σήμερα είναι η μετανάστευση. Στην καρδιά του προβλήματος πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίε της. Όμως, αν δείτε τις ειρηνευτικές ας πούμε, συμφωνίες στο Μάλι, θα δείτε ε, ότι εκεί ε, θα μπορούμε με αυτό το εργολείο πολύ πιο γρήγορα να αντιμετωπίσουμε προγράμματα που θα δείξουν τα αποτελέσματα της ειρήνης. Για τον ΩΣΑ υπάρχουν ε, ε περίπου ε, 2,5 δις που δίνονται στην Ένωση της, των Κρατών της Δυτικής Αφρικής την Επιχειρησιακή Επιτροπή του Trust Fund, που δεν έχει βέβαια δικαίωμα ψήφου ως δωρητής, διότι ο οικονομικός κανονισμός δεν το ε, επιτρέπει. Όμως, ε, ε, από τις επαφές που είχαμε μαζί τους πριν δύο εβδομάδες, μας διασφάλισαν ότι οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το Trust Fund συνδέονται με το ε, που συνδέονται με, αυτό το, με όλες τις δράσεις που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη στην περιφέρεια αυτή. Είναι 200 εκατομμύρια λοιπόν το ποσό διορθώνω. Είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν θα είναι ανταγωνιστής στην Αφρικανική Ένωση και στο εργαλείο για την ε, ειρήνη στην Αφρική, το African Peace Facility, είναι ένα ταμείο που στην ουσία θεσπίστηκε ως ε, αντικατάσταση των διμερών ε, επαφών και της βοήθειας που δίνεται σε διμερές επίπεδο και θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία τα ενδεικτικά εθνικά προγράμματα ε, που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία απασχόλησης, ε, για παράδειγμα, ή με την μετανάσταση ε, έχει μπει και το θέμα αυτό του Ταμείου. Είναι λοιπόν μια συμπληρωματικότητα που θέλουμε να δώσουμε και μια ευελιξία στη λήψη αποφάσεων. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα γι' αυτό, αλλά μπορώ να σας διασφαλίσω ότι ο σεβασμός του κώδικα ΝΤΑΚ είναι μία από τις ε, προτεραιότητάς μας στην ε, Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ. Ωραία. Θα, σας, ε, θα τα πούμε και αργότερα. Πρέπει να, Πρέπει να παρουσιάσω τη θέση του συναδέλφου μου Αρνελίτς, ο οποίος απουσιάζει. Είναι σκιώδης εισηγητής. Περίμενα να πάρω το λόγο και συνειδητοποίησα ότι μάλλον δεν ξέρατε ότι εγώ έπρεπε να παρέμβω εκ μέρου του. Θα προτείνω το εξή, λέει ο πρόεδρο. Επειδή κλείσαμε τι παρεμβάσει. Ε, μίλησε ο κύριο Ενρίκε Γκερέρο και νομίζω ότι εξέφραζε την άποψη των σοσιαλιστών. Είναι μια πρώτη συζήτηση ούτω ή άλλω. Θα κάνουμε και μια άλλη συζήτηση, ε, δεύτερη συζήτηση με κείμενο σε δύο εβδομάδε. Σα ε, πειράζει να παραιτηθείτε από το δικαίωμα λόγου και να το πείτε στην Ανλή γιατί έγινε, έγιναν πολλές παρεμβάσεις και είναι λιγάκι αργά να πάρετε τώρα το λόγο. Ιγνάσιο, θα έχουμε την έκθεσή σου σε δύο εβδομάδες. Αν θες να πεις κάτι πολύ σύντομα. Ναι, ταχύτατος. Ευχαριστώ όλους για την παρέμβαση. Για τις παρατηρήσεις. Είμαστε όλοι μέλη αυτής της Επιτροπής. Και μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη, φυσικά. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα εργαλείο το οποίο θα παίρνει κονδύλια από την αναπτυξιακή βοήθεια και θα τα βάζει, θα τα βάζει αλλού. Υπάρχει συνένεση εδώ. Ελπίζω να συνεργαστούμε, ούτω ώστε να έχουμε μια ισχυρή θέση, έτσι ως κοινοβούλιο, και να τονίσουμε την πτυχή ε, του συστήματος της παρακολούθησης, που θα είναι ο τοποτηρητής του Ταμείου. Συμφωνώ λίγο πολύ με όλες τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και ένα επιπλέον εργαλείο, δηλαδή αυτό να είναι επιπλέον εργαλείο, τόσο ώστε να έχει προστιθέμενη αξία, κάτι που ενισχύει την ε, σημασία της Αναπτυξιακής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι κάτι το οποίο απλώς μετακινεί χρήματα από την ανάπτυξη και τα βάζει αλλού στην ασφάλεια, α πούμε. Ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε, συνάδελφοι, όταν θα έχουμε την έκθεση σε μια-δυο εβδομάδε. Ευχαριστούμε και τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Τώρα έχουμε ψηφοφορίε που πρέπει να αρχίσουν 11.30 το αργότερο. Λοιπόν, κοιτάζουμε την επίσημη ανεπτυξιακή βοήθεια και την, ε, ε, τον ορισμό της. Υπάρχει η συνεδρίαση της Επιτροπής Ντάκτου αύριο για το θέμα αυτό, για την αναθεώρηση του προσδιορισμού της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και η υπεύθυνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΠΚΟ δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Ε, δεν ήρθε η ίδια λοιπόν γιατί ετοιμάζεται για την αυριανή συνεδρίαση. Ο συναδελφό τη Ζερόμ Λερουά θα μα ενημερώσει για το τι θα συμβεί αύριο στο Παρίσι. Ζερόμ, έχετε το λόγο. Σαντάλ, μάλλον. Συγγνώμη. Ε, ευχαριστώ, Λίντα. Όπω ξέρετε, η Επιτροπή ΝΤΑΚ του αναθεωρεί το στατιστικό τη σύστημα για την καταμέτρηση τη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Υπάρχουν τέσσερι βασικέ τάσει εδώ και μία επιπλέον που θα ήθελα να αναπτύξω. Καθώ όλο ο ο κ. Γκέρεν έθεσε το θέμα. Θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να απαντήσω. Η πρώτη τάση είναι ο των οδηγιών για την ειρήνη και την ε, ασφάλεια είναι θέματα που τα έχουμε δείξει και σε προηγούμενες συζητήσεις. Δεύτερη, η πρόταση να δούμε το κόστος για τους δωρητές εσωτερικώς, όπως για τους πρόσφυγες, για να έχουμε έναν σαφέστερο και διαφανέστερο τρόπο και πιο ακριβή για εργαλείο που ονομάζεται Total Official Support for Sustainable Development, όλη η επίσημη βοήθεια για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. ΤΑΦ, κάτι που θα συμπληρώσει την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και ο συνάδελφος Ζερόμ θα το αναπτύξει και τέλος πώς θα μετράμε και τις συμβολές των εργαλείων του ιδιωτικού τομέα. Δεύτερος γύρος συζητήσεων έχει γίνει μετά τις συμφωνίες του 2014 για τα κρατικά δάνεια. Το πρώτο σημείο είναι η ειρήνη και η ασφάλεια. Για τη συμφωνία του 2014 HLM ορίζει την επιφάνεια που εφάπτονται η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια με τα υπόλοιπα. Θα πρέπει η Επιτροπή ΝΤΑΚ λοιπόν να κοιτάξει πώς ακριβώς θα αποσαφηνίσει τις οδηγίες για την ασφάλεια και την ειρήνη. Μετά από ένα ολόκληρο χρόνο συζητήσεων Υπάρχει ακόμη μεγάλη ε, διαφορά απόψεων μεταξύ των διαφορών μελών του ΝΤΑΚ. Ο Βέλγος Πίτερ Μορ κλήθηκε να συνθέσει μια ομάδα για να προσπαθήσει να βρει μια συμβαστική λύση σχετικά. Έχουν γίνει λοιπόν συζητήσεις με υψηλούς εκπροσώπους των διαφόρων υπουργείων που ασχολούνται με το θέμα αυτό, το μέτρηση της επίσημης συναπτυξικής βοήθειας στα κάτι μέλη και έχουν βρει συμφωνία. Τη βρήκαν την Δευτέρα. Η νέα επικυροποιημένη οδηγία για τις αιτήσει ασύλου θέλουμε να εγκριθεί στο HLM αύριο και μεθαύριο. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες συνομιλίε για την ειρήνη και την ε, ε, ασφάλεια και η Επιτροπή μας συζητάζει με τους υπευθύνους για να δει τους, ε, το στόχο της χιλιατίας 16 και τον άλληλο συσχετισμό της ανεπίσημης αντεξικής βοήθειας με αυτό αυτό που πέτυχαν οι Βέλγοι στη βασική λύση είναι να βεβαιωθούν ότι η επίσημη αναπτυξική βοήθεια για την α, ειρήνη και την σταθερότητα σε αυτόν τον τομέα πρέπει ακόμη να περάσει το τεστ. Ε, αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες και έχει να κάνει με την ανάπτυξη χώρας στην οποία θα δώσουμε την επίσημη αναπτυξική βοήθεια. Επίσης, έχουμε δεσμευτεί να αποσαφηνίσουμε το ρόλο των στρατιωτών και της χωροφυλακής των δυνάμεων που εργάζονται στα Υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών. Πάντοτε όμως θέλουμε να διασφαλίζουμε ότι οι δυνάμεις αυτές χρησιμοποιούνται περισσότερο όταν οι πολίτες δεν είναι σε θέση να φέρουν εις πέρα στι δράσεις. Μετά ε, με την ε, με την παρακολούθηση των υπευθύνων και με διάφορα εχέγγυα. Το ίδιο έχει γίνει Ακούγεται για τα γενεσιουργά αίτια. Για τα γενεσιουργά αίτια της τρομοκρατίας. Όπου Πρέπει να χρηματοδοτηθούν άμεσα μέτρα αναθέτησης και μυστικές υπηρεσίες, αλλά θα έπρεπε να χρηματοδοτήσουμε και αυτές τις προσπάθειες καταπολέμησης των γενεσιουργών αιτίων. Το δεύτερο ζήτημα που έχει προκύψει τους τελευταίους μήνες λόγω της κρίσης των προσφύγων στην γειτονία μας και στην Ευρώπη είναι το κόστος που αντιμετωπίζουν οι δωρητές εσωτερικώς. Η DAC του ΩΣΑ έρευνα κατά πόσο οι οδηγίες αυτές πρέπει να επικαιροποιηθούν ή να αποσαφινιστούν και απέστειλε το μετολόγιο στα κράτη-μέλη. Πρόκειται για έναν τομέα όπου η τωρινή κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη και υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των κρατών μελών. Ξανακετάζουν λοιπόν τις οδηγίες τους για την επίσημη ανάπτυξη και βοήθεια και τις ειδικέ οδηγίες για τους πρόσφυγες στις χώρες υποδοχής. Θα μπορούσαν οι πρώτοι μήνες να μετράνε ως επίσημη ανάπτυξη και βοήθεια και μετά οι υπόλοιποι 12 να δούμε πώς θα χρησιμεύσουν για την επανένταξη των προσφύγων αυτών στη χώρα της, ε, στην οικονομία της χώρας υποδοχής, για την επανεγκατάσταση ενδεχομένω όπω έχουν υπάρξει και να δούμε ποια θα θεωρηθούν ODA και ποια όχι. Ε, η απέλαση των προσφύγων προφανώς δεν είναι ε, επίσημη αναπτυξική βοήθεια. Κάθε μέλος της Επιτροπής DAC πρέπει να αποφασίσει ποια ε, κόστη θα καταγράφει σε επίπεδο DAC Και υπάρχει μεγάλη ε, διακύμανση στο πώς αυτά εφαρμόζονται Πάντως, ως κράτη-μέλη βλέπουμε ότι για την ώρα δεν έχει καταγράψει κανείς το κόστος ως επίσημη αναπτύξη και βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να ε, οδηγήσει σε περισσότερο ακριβή και διαφανή καταγραφή της επίσημης ε, αναπτυξικής βοήθειας. Όμως είναι λίγο αμφίβολο το κατά πόσο θα είναι χρήσιμη επικυροποίηση τώρα, εν μέσω μια κρίσης που σοβεί και εφόσον δεν έχουν όλη την απαραίτητη ψυχραιμία. Θα πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν την απαραίτητη συνένωση, να δούμε αν έχουμε χρόνο. Και όλοι παραδέχονται ότι όσοι υπάρχουν στην οδηγία είναι καλά, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να είμαστε πιο διαφανείς στην υλοποίηση μεταξύ των μελών της ΝΤΑΚ. Ο κύριος Γκέρενς έθεσε μια ερώτηση και θα ήθελα να την απαντήσω. Η ερώτηση ήταν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει το συνολικό ποσό επίσημης αναπτυξικής βοήθειας που πανέφτει το 2015 από τα κράτη-μέλη εσωτερικός ε, για την κάλυψη του κόστου των προσφύγων ε, σε αυτό το διάστημα. Δεν έχουμε τους αριθμούς για την επίσημη και βοήθεια στις αρχές του, για το 2015 και στις αρχές του 2016. Έχουμε μόνο τα προκαταρκτικά αριθμητικά στοιχεία αυτή τη στιγμή από τα κράτη-μέλη της ΝΤΑΚ και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι μέλη της ΝΤΑΚ. Όμως φροντίζουμε να υπάρξει καταγραφή και θα κοιτάξουμε να καταγράψουμε τα πάντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατη μέλη της. Απλώς έχουμε έναν λεπτομερέστερο υπολογισμό για το 2015 αντί για το 2016. Αυτό μπορώ να σας πω λοιπόν είναι για το 2014 τι έγινε. Για το 2013 υπήρξαν συγκεκριμένοι αριθμοί και είδαμε η αλλαγή της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας να έχουν αλλάξει πολύ σχετικώς από το 2014. Δύο δεν υπέβαλαν και τα πλήρη στοιχεία. Πάντως αυτό που μας δείχνουν οι αριθμοί DAC είναι ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρουν 31 δις κόστους εσωτερικός για το δωρητή 3,31 δις ε, ως αύξηση 1,47 ε, δις από το 2013 τις τιμές του 2013 Αυτές οι δαπάνες είναι 5-6% της συνολικής επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 και οι συγκεκριμένε δαπάνες έγιναν στο πλαίσιο της αύξησης, στο σύνολο της αύξησης της ODA όπως καταγράφηκε από τα κράτη-μέλη το 2014. Οπότε συνολική επίσημη τεξική βοήθεια έφτασε τα 2,36 δις ευρώ μεταξύ 2013-2014 στην αύξησή της. Δηλαδή 59,236 εκατομμύρια 59 δις 236 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρξε αύξηση του κόστους κάλυψης των προσφύγων, αλλά υπήρξε και αύξηση στο ποσό. Στις χώρες, αυτές τα ποσά που κατευθύνθηκαν προς τις χώρες εταίρους. Θα κοιτάξουμε προσεκτικά τους αριθμούς που θα μας στείλουν τα μέλη, όμως λαμβάνουμε βεβαιώσεις ότι πάλι υπήρξε άκρηση της ODA. Και έχουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία καταγραφή στοιχείων μεταξύ κρατών μελών. Η Γερμανία δεν υποβάλλει καθόλου στοιχεία. Δεν συμπληρώνει τα στοιχεία αυτά του εσωτερικού για το δωρητή. Ενώ άλλες χώρες ναι. Ε, είναι πολύ διαφορετικό το πνεύμα λοιπόν που ακολουθεί ο καθένα. Αυτό ελπίζω ότι σα δίνει την απαραίτητη απάντηση και να δώσω το λόγο στον Ζωγόμ για να μα καλύψει υπόλοιπου τομεί. Ευχαριστώ, Σαντάλ. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να ολοκληρώσω το πλαίσιο. Πρώτον, εξυγχρονισμό των εργαλείων προς τον ιδιωτικό τομέα και το TOSST. Να ξεκινήσουμε τον ιδιωτικό τομέα προσπαθούμε να εξυγχρονίσουμε τα μέτρα δημόσιας βοήθειας για την αναπτυξιακή βοήθεια και κυρίως να λάβουμε υπόψη όλα τα εργαλεία που δεν είναι δωρές. Δηλαδή δάνεια, εγγυήσεις είναι στην πραγματικότητα και τις επενδύσεις ε, σε μετοχές, equity. Δηλαδή, το διακύβευμα είναι να δούμε τι εργαλεία έχουμε εκτός από τις δωρεές, ε, δημόσιας, δημόσια βοήθεια και η σημασία τους είναι αυξανόμενη. Το 2014 τον ΤΑΚ συνεδρίασε και υπήρξε συνένεση για τα εργαλεία που δεν ήταν δωρεές που αφορούσαν ε, τα κράτη, τις περιφέρειες και τους δήμους και κοινότητες. Ο άξονας, ο βασικός της συμφωνίας του 2014 είναι ότι μετρήσαμε τις άδειε των εργαλείων αυτών και ε, μετρήσαμε το grant equivalent, δηλαδή, δηλαδή για τα δάνεια ε, λαμβάνουμε υπόψη τη διάρκεια αποπληρωμής, τα επιτόκια κτλ. Και αυτό το ισοδύναμο δωρεάς, σε δωρεάς ήταν την, βοήθεια, τη δημόσια βοήθεια για τα δάνεια, τις εγγυήσεις και τις μετοχές. Η συμφωνία του 2014 κάλυπτε μόνο τα δάνεια προς, τον, προς το δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε ε, με συμπληρωματικά κονδύλια με δάνεια στον ιδιωτικό τομέα. Το διακύβευμα λοιπόν της συνεδρίασης της αυριανής είναι να έχουμε τις ίδιες, ε, την ίδια συμφωνία για ε, μέτρα προς την, τον ιδιωτικό τομέα. Ε, ε δάνεια, εγγύησεις και μετοχές η βασική αρχή της συμφωνίας είναι ίδια. Δηλαδή ότι ο χρυσό κανόνα τη της δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια είναι το ισοδύναμο ε, δανείου. Ποιο επηρεάζεται, οι μεγάλε χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε, CDC και τα λοιπά τη Γαλλία, η Κομισιόν δεν δίνει δάνεια. Δηλαδή, εμεί δεν επηρεαζόμαστε σε ό,τι αφορά τα εργαλεία αυτά, αλλά η ΜΠΕΗ έχει στο χαρτοφυλάκιό τη κάποια δάνεια ε, η Ευρωπαϊκή δηλαδή, Τράπεζα Επενδύσεων επηρεάζεται από αυτόν τον εξχρονισμό. Είναι πολύ δύσκολη η συνένεση, αλλά αναπτύσσεται γύρω από δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Μία θεσμική και μία ε, εργαλειακή. Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας ήταν πολύ διαιρεμένη ανάμεσα στις δύο τάσεις. Η θεσμική ε, θεωρεί ότι η κεφαλαιοποίηση ε, μιας, ενός εγκρήματος λαμβάνει υπόψη στην ε, δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια. Η άλλη θέλει να μετρήσει συγκεκριμένα με ε, ισοδύναμα δωρεών ε, τι, δίνει κάθε, τι δίνουμε με κάθε δάνειο, κάθε εγγύηση κτλ. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, είμαστε κοντά σε μια συνένεση γύρω από μια διτή λύση όπου τα κράτη-μέλη του ΝΤΑΚ θα επιλέξουν την προσέγγιση που θέλουν και αυτή τη στιγμή επιλέξουν τη συγκεκριμένη, θα κλειδώσουν αυτή την προσέγγιση για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα κινηθούν σε αυτήν μέσα. Οι αρχές είναι ίδιες για την εργαλειακή λύση, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε το ισοδύναμο δωρεάς ως ε, μέτρο για το παρεχόμενο ποσό και το σύστημα θα είναι ισοδύναμο με αυτό που χρησιμοποίησαμε περίπου για το δημόσιο τομέα, με μία διαφορά όμως, ότι δεν έχουμε κατόφλι παραχώρησης, γιατί ο κίνδυνος υπερχρέωσης ε, του ιδιωτικού τομέα ε, είναι σχεδόν μηδενικός. Αυτή είναι η κατάσταση των διαπραγματεύσεων για μας. Εμείς υποστηρίζουμε μία συνενετική προσέγγιση και μία συμφωνία για αύριο. Το διακύβευμα είναι να κρατήσουμε αυτή τη δημόσια ε, αναπτυξιακή βοήθεια και να, μπορέσουμε, και να μπορέσει αυτό που, ε, αυτό που επιλέξουμε να αντέξει σε ένα σοβαρό έλεγχο από εξωτερικούς ελεκτές Για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι έχουμε διωγγώσει τεχνητά το ποσό της αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτό μας απασχολεί όλος ιδιαιτέρως. Αυτά λοιπόν για τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα θα περάσω <clears throat> σε έναν άλλο τομέα το TOST. Total Official Support for Sustainable uh, Development. Είναι ένα εργαλείο υποτίθεται συμπληρωματικό για να δούμε τι ροέ ε, αναπτυξιακή βοήθεια δίνουμε που δεν καλύπτονται από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Είδαμε ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια κάλυπτε ένα ουσιαστικό τμήμα δημόσιας βοήθειας το TOSSD λαμβάνει υπόψη όμως όλους τους τομείς που ξεχνάμε συχνά και ε, τα δημόσια αγαθά, ας πούμε αυτό που λέμε δημόσια αγαθά, τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα που κινητοποιείται μέσω μεικτών επιχειρήσεων και την, ε, το pay security και άλλους τομείς που αυτή τη στιγμή δεν αναφέρονται καθόλου στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Η Κομισιόν έκανε ένα πιλωτικό πρόγραμμα ε, για να δει μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε με αυτούς τους νέους δείκτες και συμπεράναμε ότι ο ορισμός ε, του πλαισίου είναι σημαντικό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συνένεση σε αυτό το τομέα και σε ό,τι μας αφορούσε ο όγκος που αναφέρεται ε, ήταν περίπου συν 50% σε σχέση με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Την υποστηρίζουμε αυτούς τους δείκτες. Θαυμάσια ιδέα. Μπορούμε να βελτιώσουμε έτσι τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές οικονομικές ροές. Είναι θετικό αυτό. Δεν είναι υποκατάσταση της ε, ODA, αλλά είναι συμπληρωματικό αυτό το στοιχείο και θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τη διαφάνεια και να ξέρουμε λιγάκι περισσότερο τι γίνεται. Thank you very much. I've got two colleagues indicated so far. Ευχαριστώ. Είναι δύο συνάδελφοι που έχουν ζητήσει ως τώρα το λόγο. Κύριε Στυρ, η αναλύσα, πρώτα ο Στίβ και μετά. Λίγο γρήγορα γιατί δεν έχουμε πολύ ε, χρόνο. Ε, θα είμαι γρήγορος. Είμαι από τη Βόρεια Γερμανία και δεν μιλάμε πολύ εκεί. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε. Η κατάσταση τη επίσημη αναπτυξιακής βοήθεια στη Γερμανία είναι ένα θέμα που συζητείται αυτή τη στιγμή και αυτό που είπατε, ε, εάν ε, είναι γραμμένο στο έγγραφο, θα μπορούσα να το πάω στη Γερμανία για περισσότερη συζήτηση και διερεύνηση. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι, συγγνώμη, ε, είμαι δυσαρεστημένος γιατί αυτή η ε, βοήθεια που θα δοθεί για τα υπεράκτα εδάφη θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πανεκατάσταση των προσφύγων. Με σοκάρει αυτό, είπατε. Πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια για την επανεγκατάσταση. Ε, μιλήσατε στον Έρικ Σαλχάιμ και τι έχει να πει αυτός γι' αυτό. Θα μας πει η Κομισιόν ήδη έχουμε τα στοιχεία για ένα χρόνο για τους επιστάμενους ε, ε, κανόνες. Ο Σάρλ Κέρνς και μετά η Ανελίσσα. Να είστε σύντομο Σάρλ. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι το ε, θέμα που αναφέρετε, που είναι στο σημείο 19 της ημερήσιας διάταξης ε, μόλις αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ που απαντήσατε με εξαιρετικό τρόπο σε όλο αυτό. Ε, το ότι δεν ικανοποιούμαστε σε όλα τα σημεία είναι ε, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει ένα σύστημα και η ηλεκτρονική επικοινωνία που χρειάζεται πολύ χρόνο. Πρέπει να φτάσουμε στο 2016 στο τέλος για να έχουμε τα αποτελέσματα του 2015 και να μπορούμε να ε, δώσουμε στοιχεία για τα εξαμήνα για τις ε, ωφέλειες, τα κέρδη. Τώρα για τα στοιχεία που αναφέρατε είναι ένα εργαλείο πολύ ουσιώδους σημασίας. Πρέπει πρώτα αυτά να είμαστε σε επαγρύπνηση για να μπορεί η βοήθεια να δίνεται με τον σωστό τρόπο και πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται και με τα κονδύλια που είναι για την υποδοχή των προσφύγων. Είπατε ότι αυτό θα είναι μόνο τους δύο πρώτους μήνες, ότι αυτοί λαμβάνονται μόνο υπόψη. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Πρέπει παρόλα αυτά να δούμε εάν αυτό βοηθά την ανάπτυξη ή είναι αντιπαραγωγικό. Αν δούμε όλες τις χώρες ε, υπό ανάπτυξη, ε, αυτές Ε, με όλα αυτά που λαμβάνουν και με τη μετανάστευση που έχουμε βλέπουμε ότι δεν συμβάλλουμε στην ανάπτυξή τους αλλά στο αντίθετο μάλλον. Άρα χρειαζόμαστε ένα αναλυτικό κατάλογο με τα κόστη που έχουν δώσει τα κράτη-μέλη για τους πρόσφυγες ε, κάτω από το κεφάλαιο ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Και φυσικά φαντάζομαι ότι τα σειρματοπλέγματα που βάζουν κάποιες χώρες δεν είναι και σε αυτό το κεφάλαιο. Ε, δηλαδή υποδοχή και εγκαταστάσεις να είναι εκεί και όχι τέτοια πράγματα και νομίζω ότι αυτή η δημόσια βοήθεια για την ανάπτυξη, το κομμάτι τέλος πάντων που εμείς που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ως ε, συγκυριακό ε, θα μπαίνει εκεί. Ας πούμε, τα χρήματα που δίνονται για ένα εκατομμύριο πρόσφυγες που πρέπει να υποδεχτούμε είναι και αυτά ε, συγκυριακό θέμα και είδαμε ότι η εσωτερική κατανάλωση έχει καταφέρει ε, στη Γερμανία για παράδειγμα να αντικαταστήσει και να έχει παρουσιάσει πιο θετικά το ζήτημα. Άρα ένα θέμα τελικά ε, που εφαλεί εμάς γιατί επενδύονται χρήματα την ε, υποδοχή των προσφύγων. Η κυρία Χάουτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι ε, πρέπει να συγχαρούμε την ΤΕΦΚΟ για την εσωτερική συζήτηση που είχατε με την ΕΙΑΔ. Νομίζω ότι το λιγότερο που πρέπει να περιμένουμε τώρα είναι να συμβεί αυτό που ζητάτε, η διαφάνεια των εκθέσεων, της αναφοράς των στοιχείων γιατί με τα κριτήρια της ODA στην ουσία απομακρυνόμαστε από τις αρχές της αποτελεσματικής ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους θεσμούς της θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο περισσότερο διαφανείς νομίζω. Ευχαριστώ και η Ανελίσσα. Ρωτάει. Υπάρχουν δημόσια έγγραφα διαθέσιμα που μπορεί κανείς να διαβάσει για να τα στείλουμε στους συναδέλφους. Συγγνώμη, ο Ντάφο έχει πρώτα να πει κάτι και μετά. Ναι, πολύ γρήγορα. Θα περιορίσω το σχόλιο μου στο να πω ότι προφανώς με την έγκριση της Agenda 23 και με τους ε, ε, στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης υπάρχει αυτή η ανάγκη εξυγχρονισμού της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, άρα πρέπει να κατανοήσουμε τι συνέβη στην ΔΑΚ και τον διάλογο στην ΤΕΦΚΟ και στην ΕΙΕΒ. Όλα αυτά είναι η φυσιολογική συνέπεια, το φυσικό επόμενο μετά την έγκριση της ατζέντα και πρέπει να γίνει η συζήτηση και εδώ στο σώμα. Ήθελα να κάνω αυτό το σχόλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Σαντάλ. Όσον αφορά το κόστος ε, για τους πρόσφυγες από τους δωρητές θα πρέπει να λαμβάνετε υπο... δεν πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Δυστυχώς δεν είναι λοιπόν για τα υπεράκτια κράτη. Υπάρχουν άρθρα στο ΤΑΚ στις σχετικές οδηγίες που λένε ξεκάθαρα ότι οι δαπάνες για την προσωπική προσωρινή βοήθεια στους πρόσφυγες στις χώρες ε, τους πρώτους 12 μήνες μπορεί να θεωρούνται ODA και μπορεί να δοθεί και για την μεταφορά στην χώρα προέλευσης, την προσωρινή εστίαση και στέγαση και ε, τα έξοδα μεταφοράς της χώρας προέλευσης η οικονομία της χώρας του δωρητή ε, θα πρέπει να αναλάβει κάποια ποσά που έχουν να κάνουν που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά, την απέλευση των προσφύγων σε άλλες χώρες. Οι μετανάστες επίσης πρέπει να είναι πρόσφυγες, να έχουν αυτό το καθεστώς, να μην είναι οικονομικοί μετανάστες. Αυτό ξεκαθαρίζεται. Το που μας ενδιαφέρει είναι η αναφορά του κόστους όταν θεωρείται ODA να είναι πολύ διαφανής. Αυτό είναι το κομμάτι του δικού μας ενδιαφέροντος και δεν νομίζω ότι τώρα είναι η σωστή στιγμή να αλλάξουμε αυτές τις οδηγίες υπάρχουν, τις θέλουμε να εφαρμόζονται με διαφανή τρόπο και αυτό για τη διαθεσιμότητα των στοιχείων για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Μας ενδιαφέρει οτιδήποτε θα μπορούσε να μας δείξει τι ακριβώς δαπανάτε το συντομότερο δυνατό. Δυστυχώς, τα κράτη-μέλη στέλνουν τις εκθέσεις τους στον ΤΑΚ κάποια συγκεκριμένη στιγμή και εμείς λαμβάνουμε τα στοιχεία μόλις έχουν εξεταστεί και είναι διαθέσιμα δυστυχώς. Αυτά νομίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Κοιτάξτε συνάδελφοι, θα δούμε και τι θα γίνει αύριο στη συνάντηση. Θα υπάρξουν έγγραφα και πληροφορίες Ο Ξουλχάιν θα έρθει στην Επιτροπή, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα γιατί είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής και έπρεπε να προετοιμαστεί. Ευχαριστούμε λοιπόν την Επιτροπή που ήρθε με τόσο σύντομη, ε, με τόσο βραχυπρόθεσμη ειδοποίηση στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ και τώρα συνάδελφοι περνάμε στις ψηφοφορίες. Έχουμε πολλές, αν μπορεί κάποιος να μου φέρει τον κατάλογο θα με βοηθούσε. Ξεκινάμε με το σημείο... Πρώτα απ' όλα να κάνουμε έναν έλεγχο, να δούμε αν λειτουργούν όλοι, αν λειτουργούν τα μηχανήματα όλων. Πατήστε το κουμπί. Δουλεύουν τα μηχανήματα. Okay or nerves, we can add you. It doesn't matter, nerves, We can add you in. So don't worry checking the minute. The vote is closed. Πέρας. Ωραία. Βλέπουμε ποιοι λειτουργούν. Μια χαρά. Δουλεύουν τα μηχανήματα. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Πρώτο σημείο. 8. Απαλλαγή 2014. Ταμείο Ανάπτυξης. Κύριε Φρουντζουλίτσα, έχετε κάτι να πείτε. Είστε πολύ δημοφιλής εισηγητής. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία από τον εισηγητή. Στο τέλος της, του καταλόγου υπέρ προφορική τροπολογία 1 στο τέλος του καταλόγου των ψηφοφοριών σας συμπεριλαμβάνεται. Και Στία, στο κατάλογο ψηφοφοριών του ΕΛΚ, στη σελίδα 5, έχουμε άλλη σειρά προφανώς από τη δική σας, οπότε δεν το βλέπουμε. Ωραία, να τα βρει και το ΕΛΚ και προχωρούμε. E We're voting on the discharge of... Αναπτυξιακό ταμείο, αυτό ψηφίζουμε. Εντάξει, Ντάβο. Ε, να δούμε λοιπόν αν έχουμε την ίδια... Α, έχετε δίκιο, δεν ακολουθούμε τη σειρά της ημερήσιας διάταξης. Αναπτυξιακά ταμεία. Ξαναρχίζουμε με το άλλο σημείο. Ναι. Ναι, συνάδελφοι, που να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Έχω λάθος αρρύθμιση εδώ στα έγγραφα. Έχω λάθος κατάλογο. Συνάδελφοι, ξαναρχίζουμε. Απαλλαγή για το γενικό προπολογισμό πρώτα. Γενικό προπολογισμός. προπολογισμο προπολογισμός Γενικός 2015-21-54 Να ψηφίσουμε μπλοκ τι τέσσερις πρώτε τροπολογίε. Εάν το δέχεστε ψηφίζουμε τι τέσσερι πρώτε μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την 5. Ε, Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 6. Σε χωριστά τμήματα. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα. Πέρας. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 Ποιο καταπίπτει? Η 9 καταπίπτει. Πάμε στη 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τη 10 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός 1. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 11 καταπίπτει. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θαυμάσια τροπολογία. Η 14 πάμε τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, α, το πρώτο τμήμα, υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, τη 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την έκθεση, την γνωμοδότηση μάλλον διορθώνει, όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίστε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας φοφορίας Εγκρίνεται με 22 υπέρ, 4 κατά. Αλλά έχετε και ακόμα μία έκθεση. Η έκθεση για την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου. Πού είναι ο κατάλογος μου, τον έχασα. Ο κ. Πρέντα θέλει να προτείνει να ψηφίσουμε τις τέσσερις πρώτες μαζί. Οι τέσσερις πρώτες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Έχουμε μια προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Ε, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 11 ηλεκτρονικά. Ψήσαν όλοι. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Βραχία κεφαλή με μία ψυχοϊπέρα Παραπάνω πέρασε. 12. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Αποχές. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζεται τώρα. Πέρας φοφορίας. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Εγκρίνεται η 13. Ελέγχουμε χρονικά τη 13. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δίκιο είχατε. 14. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 16.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 τη συνεργασία τους. Okay. We now move Και τώρα πάμε στο σημείο 10 για το μας στην Γρυλανδία. Δεν υπάρχει τροπολογία. Ψηφίσουμε συνολικά την έκθεση. Ψηφίσουμε τώρα ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ, μία ψήφος κατά, εγκρίνεται, ευχαριστούμε. Κύριε Κούλογλου, σας ευχαριστούμε για τη δουλειά σας. Πάμε τώρα σε μια μακρύτερη, μακρύτερο κατάλογο ψηφοφοριών, γνωμοδότηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα ε, νέο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ε, έκθεση Hayes. Έχουμε διάφορες συμβαστικές ε, σε αυτή την έκθεση. Ελπίζω να μην ε, μας πάρει πολύ χρόνο. Η πρώτη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε γιατί δεν ξέρω. Η τροπολογία 23 ψηφίζεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ολοκληρή έκθεση. Ε, ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 Μία ε, υπέρ, ε, μία αποχή. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο του ε, τους Σκιώδη, το προσωπικό που έκαναν τους συμβασμούς και έκαναν τη ζωή μας πιο εύκολη. Τώρα περνάμε σε μια πιο ουσιαστική έκθεση. Είναι η έκθεση για τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη. Ο εισηγητή είναι ο κύριο Στέβα. Θέλετε να πείτε κάτι πριν την ψηφοφορία. Να ευχαριστήσω μόνο του συναδέλφου μου για την τεράστια συνεργασία που είχαμε με όλους. Προσπάθησα να καταλάβω τη δική τους άποψη και αυτοί προσπάθησαν να καταλάβουν τη δική μου. Ευχαριστώ λοιπόν γιατί πολλές από τις συμβαστικές τροπολογίες ε, που έχουμε εδώ σε αυτό οφείλεται. Ήταν μεγάλο το ζήτημα και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βλέπω πολλές ε, ε, διατυπώσεις εδώ στις ε, τροπολογίες της συμβαστικές και από τον εισηγητή και από το προσωπικό. Ξεκινάμε με τη συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 91. Υπέρ. Κατά. Δεν ψηφίσατε. Παρακαλώ ψηφίστε συνάδελφοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ε, συμβαστική. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Όχι. 102. Ε, τροπολογία 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 102. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξω και την 103. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Όχι ακόμα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε και την 110. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται αυτή. Συμβαστική 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 118 και 19 είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. 118-119. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε την 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Άποχες. Πρέπει να ελέγξουμε και την 122. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 127. Υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται αλλά σε ελέγξουμε την 127 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 142, 43, 44 υπέρ, κατά, αποχές, Για να ελέγξουμε την 142 γιατί οι φιλελεύθεροι δεν βλέπω τι κάνουν. 142 κάνουν τη διαφορά. Άρχεται η ψηφοφορία πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική 26 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146, 147, 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149. Όχι, καταπίπτει. 150 και 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 151. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται. Συγγνώμη. 153 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε, άρχεται η ψηφοφορία, 153, ψήφισαν όλοι, πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε και την 152 γιατί δεν εγκρίθηκε η 151. 152, πάμε μία πίσω, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 152, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτεται. 153, όχι το κάνουμε. 154 και 155, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 156 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα περάσουμε στην ε, συμβαστική 19. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39, 30 ε, αλφα μάλλον. Εγκρίνεται. 169 ως 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε την 172. Έχουμε τη συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 ε, συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για να πάω την 184 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 185-86 υπέρ κατά αποχές εκρίνεται. 187 καταπίπτει καταπίπτει καταπίπτει 190-92 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ας ελέξουμε Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 194. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 196 98 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι είναι το ίδιο αλλά θα ελέγξουμε ανοίγουμε την ψηφοφορία για το 196 198 ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτεται είναι πλειοψηφία συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 201 περιμένετε όχι 199 η, αυτή η πρόταση εκεί καταπληκτή, άρα ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, για να το ελέγξουμε. Ψήφισαν όλοι πέρας ε, της ε, ψηφοφορίας εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 201 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 211 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε το δεύτερο σημείο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Καταπίπτει. Η 212 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται νομίζω. Για να ελέγξουμε τη 212, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Συμβαστική 37, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 218 υπέρ, 200... Ε, συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη 218. Υπέρ κατά αποχές. Δεν βλέπω γιατί κάποιοι δεν ψηφίζουν. Να, να δούμε την 218 υπέρ. Συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 219. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πρώτο τμήμα της 219, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Αλλά να ελέγξουμε. Αλλά μοιάζει να υπάρχει πλειοψηφία. Οπότε πάμε στη 220 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη συμβαστική 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 248 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 249 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ας ελέγξουμε τη 249. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Όμως ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται όντω. Τροπολογία 250. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και πάλι ψηφοφορία. Συμβαστική 33, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 34, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 35, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική, όχι, συγγνώμη, τροπολογία 267. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Για να ελέγξουμε τη 267. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 268. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36. Συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 274. Από τον εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία απορρίπτεται. Συμβαστική 1 στις ιδεολογικές σκέψεις. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά πάμε στην τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 21-23 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές να την ελέγξουμε την 21 έως 23, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ωραία, εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε την 24, αλλά την 25, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26. Όχι. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27, 28, 29 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 30 με 31. Ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 32 34. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44, 45, 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορία, Απορρίπτεται. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Δεν καταπίπτει. Γιατί προηγούμενη απορρίφθηκε. απορρίφθηκε. Υπέρ της 56. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται για να την ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψήφο. 58 ως 60 υπέρ. Κατά. Θα το δούμε. Ελέγχουμε την 58 ως 60. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 61 ως 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 66 μάλλον υπέρ κατά αποχές για να την ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρασε τη ψηφοφορία απορρίπτεται. Συμβαστική υπέρ, 5 ε, ε, υπέρ, κατά, εξήντα είναι ταυτόσιμη, όχι όχι, μπερδεύτηκα, συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 2. Πάμε στη συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 76 έως 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80 όχι, 79. Είναι χωριστή. 79. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές ναι, δεν μπορώ να καταλάβω 83 άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται 84. Όχι. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές αναφορέ τι ξέχασα. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Μπορούμε να ψηφίσουμε από την 3 ως την 13. Unblock. Ομαδικά. Ναι. Όχι, δεν ψηφίζουμε μπλοκ. Δεν συμφωνούν όλοι. Τρία. Γρήγορα μπορείτε. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τέσσερα. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Πέντε. Έξι, επτά. υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Οκτώ. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Εννέα. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Δέκα. 11, ε, δώδεκα. υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Δεκατρία. υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Όχι, πρέπει να ψηφίσουμε και τη γνωμοδότηση Άφετ. Υπάρχουν σας που δεν τι ψηφίζουμε, ωραίο αυτό. Παράγραφος 4 νομίζω ότι είναι η πρώτη, έτσι. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Δεν μπορώ να καταλάβω, οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε πέρα, 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η νομοδοτηση τα ίντα, ένα-δύο πράγματα που πρέπει να ψηφιστούν. Τέσσερα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνονται. Επτά, υπέρ. Κατά. Αποχές, έλεγχος. τα. επτά, αρχική ψηφοφορία, ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. Οκτώ, τα. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστική. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικό συνάντρυφη. Μου πέσα το τηλέφωνο. Ψηφίζουμε ονομαστικά. Εψήφισαν άπαντε. Ωραία. Εγκρίνεται. 21 προς 5. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια κύριε Ντεβά. Πολύ δουλειά. Πολύς χρόνος. Σας ευχαριστούμε για όλη σας τη σκληρή δουλειά. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τις τροπολογίες της ψηφοφορίας. να πω, τελειώσαμε νωρίτερα. Να θυμίσω στους συντονιστές Να θυμίσω στους συντονιστές ότι έχουμε γεύμα με την Ολλανδία Υπουργό στις 12.30 στο Εστατήριο των Μελών. Θα σας ξαναδώ στις 3.00.